Guten Tag. Wir beginnen unsere Sitzung. Καλησπέρα σας. Αρχίζουμε τη συνεδρίασή μας για να μην περιμένει η κυρία Επίτροπος και πάρα πολύ. Υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ημερησία διάταξη. Δεν έχει παρατηρήσει εδώ αυτής. Ωραία. Σημείο 2 έγκριση των πρακτικών. Τα έχετε τα πρακτικά αυτά μπροστά σας. Ω συνήθω πρέπει να τα διαβάσετε και στο τέλος της συνεδρίας να μου πείτε αν έχετε παρατηρήσει ή όχι. Εάν όχι, εγκρίνεται. Η συνεδρίαση εγκρινεται η σε αναμεταδίδεται στην τηλεόρασή μας. Εκτός από τσεχικά, λιθονικά και εσθονικά και μελτέζικα έχουμε όλες τις άλλες γλώσσες. 16 γλώσσες όλο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αύριο δεν συνεδριάζουμε σε αυτή την αίθουσα. Αύριο για την ψηφοφορία και για την ακρόαση για τον κινηματογράφο συνεδριάζουμε στο άλλο κτίριο στο Γιάν Γιάν 4Q1 μην το ξεχάσετε αυτό και παρακαλώ να πάρετε κιόλα σας τα πράγματα που έχετε εδώ που τα χρειαζόσαστε αύριο μην αφήσετε εδώ τίποτα γιατί ίσως υπάρχει άλλη συνεδρίαση εδώ ή μπορεί να χρειαζόσετε τα έγγραφά σας για να ξέρετε τι ψηφίζετε σας παρακαλώ να πάρετε στα έγγραφά σα την ε, έκθεση για την επίσκεψη αντιπροσωπεία μα στο ΠΕΣ. Πολιτιστική πρωτεύουσα. Πάρα πολύ επιτυχής αποστολή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου και με τη Επιτροπή μα, κύριο Τέοκε, που ήταν επικεφαλή τη αντιπροσωπεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κριστιανή και την κυρία Τούλινγκ από την Γραμματεία που οργάνωσαν τα πράγματα θαυμάσια. Η αντιπροσωπεία μα είχε δυνατότητα να συζητήσει και με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό. Είχε μεγάλο αντίκτυπο στην κοινή γνώμη αυτή η επίσκεψη. Όταν πηγαίνουμε σε χώρες που δεν είμαστε πολύ συχνά, ίσως μας βλέπουν περισσότερο και αυτό χαίρομαι που η πολιτιστική πρωτεύουσα Πέτσο και η αντιπροσωπεία που πήγε επί είχε τέτοιο αντίκτυπο στον τύπο και στα ΜΜΕ γενικά. Αν έρθει τώρα η κυρία θα χαρώ. Α, εδώ είναι. yeah. the So I, uh, I have pleasure to welcome. Έχουν ευχαρίστηση να καλωσορίσω την Επίτροπο στην Επιτροπή μας εδώ. Δεν είναι βέβαια ένα μεμονωμένο και έκτακτο γεγονός, είναι συνήθες, έχουμε μια τακτική ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε διάφορα ενδιαφέροντα σημεία που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας. μόλις ε, ετοιμαζόμαστε να εγκρίνουμε το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2011, κάπου 10, 11, 12 χρόνια δεν θυμάμαι, από τότε που ξεκίνησαν πολλά προγράμματα και πραγματικά ώρα είναι να συζητήσουμε μαζί σας τις δυνατότητες που έχουμε. Και οπωσδήποτε μετά το 2014 θα έχουμε νέα προγράμματα που θα αρχίσουμε να τα συζητάμε για να έχουμε το πιο καλό πρόγραμμα που είχαμε ποτέ. Κύριε Επίτροπε, Αντρούλα, ναι, ίσως έχετε τώρα μία σύντομη, ίσως και πιο μακρά παρουσίαση και μετά μέχρι τις 4.30 θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί σας τα τρέχοντα ε, γεγονότα και άλλες ιδέες που έχετε. Uh, Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Ντόρις, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας στα πλαίσια αυτού του δομημένου διαλόγου που έχουμε τακτικά με το Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τις πολλές και πολύτιμες εκθέσεις που ολοκλήρωσε και που προετοιμάζει για τη φετινή χρονιά. Είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά το 2011 με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νέα προγράμματα και προωθώντας βεβαίως την ατζέντα για την εκπαίδευση και, ε, τον πολιτισμό. Στα εισαγωγικά μου σχόλια θα εστιάσω σε τρεις τομείς. Πρώτα απ' όλα για την νεολαία σε κίνηση, για το follow-up της Πράσινης Βίβλου για τις ε, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες και για τον αθλητισμό. Θα αρχίσω με την στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Αύριο η Κομισιόν θα εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών για το 2011. Αυτό σημαδεύει την αρχή του δρόμου που θα ακολουθήσουμε προς τους στόχους της Ευρώπης 2020 και τη στιγμή που θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τις εμβληματικέ μας πρωτοβουλίες. το βασικό μήνυμα της Ευρώπης του 2020 είναι απλό και σαφές. Αν θέλουμε να βγούμε από την κρίση με το κοινωνικό μας μοντέλο και την ε, παγκόσμια θέση μας ε, ανέπαφα, ε, πρέπει να προωθήσουμε μια έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη με την, όπου, να συμμετέχουν όλοι. Αυτό αντικατοπίζει ακριβώς το σκοπό της εκπαίδευσης της ε, ε, παιδείας και της κατάρτισης. Πρέπει να ε, το επιδιώξουμε αυτό μαζί, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την αριστεία και την ισότητα. Το πρόγραμμα Νεολαία σε που είναι η εμβληματική μου πρωτοβουλία για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, βασίζεται ακριβώ σε αυτού του δύο πυλώνε. Θέλουμε να δώσουμε στου νέου ανθρώπου ε, το δυνατότητα να υποφελθούν πλήρω από μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση. Οι, Ευρώπη πρέπει να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπορέσουν να ανταποκριθούν στι αυξανόμενε ε, ανάγκε για ειδική, ειδικέ δεξιότητε στην αγορά εργασία. Και τα πανεπιστήμια πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό. Αλλά Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η παιδεία ε, θα δώσει ευκαιρίες για όλους και θα περιορίσει τις ε, ε, ανισότητες. Γιατί για κάποιες ομάδες της κοινωνίας μας δεν είναι αρκετό να δώσουμε τα εργαλεία για την οικονομία της γνώσης, διότι ήδη εξ αρχής κάποια στρώματα είναι ήδη αποκλεισμένα. Πρέπει ενεργά να προσπαθήσουμε να τα σωματώσουμε στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και άτυπης και επίσημης. Η νεολαία στην, σε κίνηση είναι η καρδιά της Ευρώπης του 2020. Πιστεύω ότι δίνει το, την πολιτική εστίαση για την κοινή μας δουλειά σε αυτή την Επιτροπή και δίνει ε, νέα ενέργεια στις μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών στον τομέα της εκπαίδευση και τη κατάρτιση. Να σα πω με δύο λόγια πώ θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα Νεολαία σε Του χρόνου θα ξεκινήσουμε μια νέα στρατηγική πρωτοβουλία ε, σχετικά με τον εξυγχρονισμό της ανώτερης εκπαίδευση. Οι στόχοι μα είναι σαφεί. Να διευρύνουμε την πρόσβαση ε, για φοιτητέ από κάθε προέλευση και να κάθε background και να έρθουμε πιο κοντά στον ευρωπαϊκό στόχο του 40% συμμετοχή των νέων στην, ε, ε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να ε, εξασφαλίσουμε ότι οι απόφοιτοι θα έχουν ε, αποσχολήσιμες δεξιότητες και να, να αποφελθούμε πλήρως από την μεγάλη ποικιλία που έχουν να προσφέρουν τα πανεπιστήμια μας και να βρεθούμε στην παγκόσμια σκηνή, ούτω ώστε η ανώτερη εκπαίδευση της Ευρώπης να είναι συνώνυμη με την αριστεία. Να σας αναφέρω δύο πρωτοβουλίες που έχουμε υπόψη μας. Για να προωθήσουμε ε, το άνοιγμα αυτό, εξετάζουμε την δυνατότητα να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα για την χαρτογράφηση των διαφορετικών ισχυρών σημείων των πανεπιστημίων μας. Ένα τέτοιο σύστημα θα ανταποκρίνεται στην ε, ποικιλομορφία των Ευρωπαϊκών Συστημάτων της Ανώτερης Εκπαίδευσης και θα βοηθάει τους φοιτητές να κάνουν μια ε, επιλογή ε, εν πλήρη επιγνώση του από πού θέλουν να φοιτήσουν. Επίση, εξετάζουμε τη δυνατότητα δανειοδότηση των φοιτητών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο σκοπό μα είναι να προωθήσουμε την διακρατική ε, κινητικότητα των φοιτητών και να βελτιώσουμε την πρόσβαση των νέων στην ανώτερη εκπαίδευση. Θα ήθελα να επανέλθω τώρα στην ισορροπία ανάμεσα στην αριστεία και την ε, ισότητα για να γίνει, για να συμμετέχει μάλλον ο καθένας στην ανώτερη εκπαίδευση, έχουμε την ευθύνη να επενδύσουμε στα πρώτα ε, χρόνια της σχολικής ζωής. Θα προτείνω μια σύσταση στα κράτη-μέλη σχετικά με πολιτικές για την καταπολέμηση της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου. Φυσικά αυτός είναι ο δεύτερος ευρωπαϊκός μας στόχος όσον αφορά την εκπαίδευση. Να μειώσουμε την πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου σε ένα ποσοστό κάτω του 10%. Επίσης με το ίδιο πνεύμα θα προτείνω μια σύσταση για την ε, ε, άτυπη και ανεπίσημη μάθηση. Ε, εθνικά ε, συστήματα ε, προσόντων που θα πρέπει να αναγνωρίζουν δεξιότητες που αποκτώνται εκτός της επίσημης και τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρέπει οι νέοι να μπορούν να κινούνται ανάμεσα στην επαγγελματική κατάρτιση και τα πανεπιστήμια πιο εύκολα. Η διαβίου μάθηση επίσης είναι ε, η, μια αρχή που μας καθοδηγεί στις δράσεις μας αυτές. Αν σκεφτούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί μπορεί να προσθέσει αξία στις προσπάθειες των κρατών μελών, τότε είναι σαφές ότι θα πρέπει να ε, εστιάσουμε στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ε, τα προγράμματα μας πρέπει να εστιάζουν στην ε, ανάπτυξη που θα αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Υπάρχει τεράστια ε, ζήτηση, μία ζήτηση την οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με τους σημερινούς στόχους ε, και πόρους και θα πρέπει να τη διαχειριστούμε αποτελεσματικά. Του χρόνου θα έρθουμε με προτάσεις μας για την ε, επόμενη γενιά προγραμμάτων. Απευθύνω λοιπόν μια έκκληση σε εσά να είστε φιλόδοξοι σε σχέση με τα προγράμματά μας. Είμαι επίσης πεπισμένη ότι η διατήρηση ισχυρών ταυτοτήτων είναι το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή τώρα για να αυξήσουμε ε, τις εισρωές μέσω συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων, μέσω εξυγχρονισμού των στόχων ε, των προγραμμάτων, απλοποιώντας τις διαδικασίες και αναπτύσσοντας την ικανότητά τους να ε, προσελκύσουν ε, κονδύλια από, άλλους, ε, από άλλες πηγές όπως από τοπικές ή περιφερειακές αρχές. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τώρα να αναφέρω δύο πράγματα για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες πριν να έρθω στον αθλητισμό. Ε, ήταν κρίσιμη η χρονιά για ο πολιτισμό και η δημιουργική τομή στην πολιτική ατζέντα. Ο δημιουργικός ε, τομέας έχει ε, ένα ρόλο κεντρική σημασίας για την πρόθεση της καινοτομία, των δεξιοτήτων, για την πρόθεση της πολιτιστικής πολυμορφίας, εκμεταλλευόμενο όλες τις ευκαιρίε του ε, ψηφιακού ε, κόσμου. Πιστεύω ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να βοηθήσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό να δημιουργήσει βιομηχανίστη ε, βιομηχανίες κλάδους, αν θέλετε, για να γίνει η μετάβαση σε, ψηφιακές πλατφόρμες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτά με έναν τρόπο ευφυή e, που θα αναγνωρίζει που οι αγορές δεν μπορούν να λειτουργήσουν και που οι πολιτιστικοί παράγοντες και φορείς χρειάζονται δημόσια υποστήριξη. Αυτό ε, απαιτεί τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για το copyright που προωθεί την πολιστική ε, πολυμορφία και ε, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα ε, σε όλους τους πολιστικούς τομείς. Στον οπτικοακουστικό τομέα θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την κίνηση προς ε, πανευρωπαϊκές άδειες για κατόχους δικαιωμάτων που τις θέλουν, ενώ παράλληλα θα σεβόμαστε τη βασική αρχή της συμβατικής ελευθερίας. Του χρόνου θα ασχοληθούμε με τα θέματα που προέκυψαν από τη διαβούλευση για την ε, πράσινη ε, βίβλο με μια νέα ανακοίνωση. Ο σκοπός μας είναι να προωθήσουμε και να κάνουμε να ανθίσει ένα περιβάλλον όπου μπορούν να ανθίσουν οι δημιουργοί τομεί, κάνοντας πιο εύκολη την πρόσβαση στην ε, χρηματοδότηση, παρακολουθώντας τις ανάγκες για νέες δεξιότητες και ενσωματώνοντας τις τις βιομηχανίες αυτές σε περιφερειακές αναπτυξιακέ στρατηγικές και επίσης δημιουργώντας δημιουργικέ δημιουργικές σχέσει σχέσεις ανάμεσα στην ε, παιδεία, τι επιχειρήσει και τους ε, δημόσιου ε, φορείς. Πρόκειται για έναν ζωντανό δημιουργικό κλάδο που θα ενσωματώσει, θα, θα, ενδυναμώσει την πολιτική πολυμορφία της Ευρώπης. Επίσης θα έχουμε ένα σχήμα υποστήριξης για τον κινηματογράφο που θα περνάει στην ε, ψηφιακή τεχνολογία. Αυτή η υποστήριξη είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν αφήσουμε τους κινηματογράφους να κλείσουν γιατί είναι πολύ δύσκολη η μετάβασή τους στην ψηφιακή τεχνολογία, τότε θα έχουμε σε κίνδυνο την πολιτιστική μας πολυμορφία. Και αυτό είναι αυτό που εννοούμε ε, όταν λέμε ότι θα προωθήσουμε το δημόσιο συμφέρον στον πολιτισμό. Οι αγορές από μόνες τους δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά χρειάζεται ε, δημόσια υποστήριξη. Και μια και μιλάμε για την ευρωπαϊκή ταυτότητα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε για την ευρωπαϊκή ετικέτα, την ετικέτα ευρωπαϊκής κληρονομιάς, την οποία θα ψηφίσετε αύριο, αν δεν κάνω λάθος, και ιδιαίτερα την κυρία Παγιοντέλη. Ευχαριστώ όλους ιδιαίτερους. Ε, ελπίζω ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία μας ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό κείμενο. Ας συνεργαστούμε ούτως ώστε η ετικέτα αυτή να κερδίσει την ε, ε, αξιοπιστία και το κύρος που της αξίζει. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα παρουσιάσω φέτος μια ανακοίνωση για τον αθλητισμό. Μια ανακοίνωση. <laughs> ναι, ναι, ανακοίνωση, το κατάλαβα. Ε, που θα προσδιορίζει την πολιτική πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευρωπαϊκή και εθνική δράση για την προώθηση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού ρόλου του αθλητισμού. Η ανακοίνωσή μα θα δίνει κατευθυντήρε γραμμέ και υποστήριξη στο αθλητικό κίνημα σε όλα τα επίπεδα. Στο ε, ερασιτεχνικό και στο επαγγελματικό επίπεδο και θα ε, δείξει την δέσμευσή μας να ενισχύσουμε το διάλογο μαζί τους. Ε, δυστυχώς, ε, δημοσιονομικοί περιορισμοί και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2012. Πιστεύω όμως ότι είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε τη μελλοντική μας πολιτική με πρακτικές ενέργειες στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συνεχίσουμε τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που ήδη ε, ξεκίνησαν παραπάνω από 30 διακρατικά project τα τελευταία δύο χρόνια. Ε, ο προϋπολογισμός του 2011, για τον οποίο πολεμήσατε τόσο σκληρά, θα χρηματοδοτήσει δράσεις το 2012 και κατά πάσα πιθανότητα και μετά από αυτή τη χρονιά. Θα είμαστε λοιπόν έτσι σε θέση, ε, κατόπιν αυτού, να αξιολογήσουμε τις δράσεις σε περισσότερους από 12 τομείς της πολιτικής αθλητισμού και να κάνουμε μια ε, σε βάθος ε, αξιολόγηση αντικτύπου αυτό θα μας δώσει μια στέρεα βάση στην οποία να βασίσουμε την μελλοντική μας ε, δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκίνησα μιλώντας για τους προϋπολογισμούς. Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας πόσο ευγνώμων είμαι για την υποστήριξη αυτής της Επιτροπής και τις προσωπικές σας προσπάθειες να αντισταθείτε στις περικοπές του προϋπολογισμού που προτάθηκαν από το Συμβούλιο για το 2011. Παράλληλα με τις προετοιμασίες μας για τα νέα προγράμματα, ε, η ενδιάμεση αναθεώρηση του προπολογισμού έχει ήδη προκαλέσει μια ε, πολύ έντονη συζήτηση για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, μαζί έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να μεταρρυθμίσουμε τον προϋπολογισμό μας ώστε να υπηρετεί όπως χρειάζεται τους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη του 2020 έχει στην καρδιά της, ε, στους στόχους της, την εκπαίδευση. Τώρα χρειάζεται ένας ε, προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να ανταποκρίνεται σε αυτές τις προτεραιότητες. Είναι η εκπαίδευση, κυρίες και κύριοι, που θα βοηθήσει να μπει η Ευρώπη στο δρόμο για μια έξυπνη ανάπτυξη με την συμμετοχή όλων. Η εκπαίδευση θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε κάποιες από τις πιο βαθιές ανισότητες της κοινωνίας μας. Της κοινωνίας μας και είναι η εκπαίδευση, είναι η παιδεία αυτή που θα μπορέσει ε, να ε, οδηγήσει στην ε, ολοκλήρωση των διαφόρων κοινοτήτων και κοινωνιών σε μια περίοδο έντασης των κοινωνικών αναταραχών. Ε, με, αυτούς, ε, με αυτές τις σκέψεις ε, ελπίζω ότι θα συνεχιστεί η οικοδομητική συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Έχετε δίκιο. Η παιδεία είναι το α και το ω. Και εδώ και στις πατρίδες μας και την Κυριακή και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή που εκείνοι που εργάζονται στα ε, ε, στα Υπουργεία ξεχνάνε πόσο σημαντικό είναι. Τώρα θα περάσω στα γερμανικά πάντα και θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους γιατί αν δεν μιλάω γερμανικά θα με μαλώσουν στη Γερμανία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ακούσαμε, αυτοί είναι οι κύριοι πυλώνες τα κύρια θέματα είναι η ανώτερη εκπαίδευση και εκείνοι που εγκαταλείπουν τη σχολική του εκπαίδευση προώρα. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να δράσει η Κομισιόν εδώ. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει οπωσδήποτε η διαδικασία της Μπολόνια να ε, εστιαστεί καλύτερα στις ιδέες της Κομισιόν, αλλιώς δεν μπορούμε ποτέ να επιτύχουμε αυτό που θέλουμε. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι ακριβώ ότι με το θέμα της, του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ε, μπορούμε να περάσουμε ένα σημαντικό τμήμα της εργασίας μας στο επίκεντρο της ε, προσοχής των πολιτών. Ε, από στο Βερολίνο έχω να συμμετάσχω σε ένα συνέδριο που έχει τον τίτλο Culture Invest, επένδυση στον πολιτισμό. Και έτσι καταλαβαίνουν πολύ ότι αυτό θα πρέπει να είναι στο αυτό στο οποίο θα πρέπει να βασιστούμε. Εγώ δεν έχω σας υποβάλω ερωτήσεις, κύριε Επιτροπέ. Θα ήθελα οι συνάδελφοι να σα υποβάλουν ερωτήσει. Ο κύριο Μιγάλσκι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο. Θυμάμαι ότι σας συνάντησα όταν είχατε εκλεγεί στο αξίωμα αυτό ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία μας τότε. Σας είχα κάνει κάποιες ερωτήσεις για τα μέτρα και για τις πρωτοβουλίες τις οποίες ε, θα υιοθετούσατε σε σχέση με τις ε, χώρες που είναι ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξή Του χρόνου προβλέπετε κάποιες νέες, και παραλαμβάνω τη λέξη, νέες πρωτοβουλίες, δηλαδή πρωτοβουλίες που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις έξι χώρες που είναι στο πρόγραμμα για την σχέση την εταιρική με την Ανατολή. Μπορείτε να διευκρινίσετε μερικά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, αυτό το οποίο θα με ενδιέφερε θα ήταν να ακούσω κάποια πράγματα για τα σχέδια της Επιτροπής ε, σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Δεν είναι και τόσο ρόδινη κατάσταση, ε, φοβούμε, σε σχέση με αυτά που μας είπατε. διότι δεν υπάρχει ένα κοινοτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης ε, του αθλητισμού μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου που υποτίθεται ότι θα συνόδευε την ανακοίνωση για τον αντίκτυπο της συνθήκης της Λισαβόνας. Πότε αναμένεται να δημοσιευθεί η έκθεση σχετική και δεύτερο ερώτημα πρόκειται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει τον αθλητισμό στα ήδη φυστάμενα προγράμματα χρηματοδότησης, διαβίου, μάθηση, ε, η πολίτες για, για την Ευρώπη, όλα τα σχετικά προγράμματα. έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι χρηματοοικονομικοί όροι για κάποιες αθλητικές εκδηλώσεις ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Ίσως για φέτος ή για το ε, ερχόμενο έτος. Η κυρία Χαίρομαι που σας βλέπω κυρία Βασιλείου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα μιλήσω ελληνικά για να με μαλώσουν οι δικοί μου συνάδελφοι και για να καταλάβει και η κυρία Βασιλείου, μια και μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ε, θα αναφερθώ μόνο σύντομα στο πρώτο κομμάτι της ε, εισήγησή σα, που αφορά στον εξυγχρονισμό της, ε, ανώτερης της, της πανεπιστημιακής Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ε, την φθήνουσα πορεία των ανθρωπιστικών σπουδών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, δεδομένου ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές συνδέονται άμεσα με την κουλτούρα της Ευρώπης, με τον πολιτισμό της Ευρώπης, ε, υπάρχουν τρόποι, έχετε σκεφτεί, προγραμματίζετε να αναζητήσετε προκειμένου να ενισχυθούν με κάποιο τρόπο οι ανθρωπιστικές σπουδές στα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ξιότιμη κυρία Επίτροπε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να χαιρετήσω την απόφαση σε σχέση με το επόμενο έτος. Είπατε ότι σχεδιάστε να συντάξετε ένα νέο πρόγραμμα για τον εξυγχρονισμό της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια θα συνεχίσετε τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας της Μπολόνια. Βέβαια θεωρώ ότι αυτό έρχεται με κάποια καθυστέρηση. Θα έπρεπε ήδη να είχε υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό για να αποφύγουμε το κενό μεταξύ της ολοκλήρωσης της πρώτης δεκαετίας της Μπολόνιας και τη συνέχιση των προσπαθειών μας. Είμαι πεπισμένος ότι η φιλοσοφία θα παραμείνει ίδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εν γέννη, θα πρέπει να στηρίξουν ε, περαιτέρω ορισμένα προγράμματα. Στι δηλώσει, σα μεταξύ άλλων αναφέρατε ότι είστε ικανοποιημένοι με <clears throat> την προηγούμενη δεκαετία και τι μεταρρυθμίσει στον τομέα τη ανώτερη εκπαίδευση. Είπατε ότι η διακήρυξη τη Μπολόνια έχει εμπνεύσει διάφορε χώρε ε, στο να υιοθετήσουν ε, σύγχρονε πρακτικές και προσεγγίσεις. Είπατε ότι πολλά έχουν γίνει, αναφέρατε όμω ότι μένει ακόμη να γίνουν πολλά και δει στον τομέα τη ανώτερη εκπαίδευση, εάν θέλουμε να πετύχουμε κάποιου ε, ουσιώδει στόχου. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από εσά σε ποιου πυλώνε θα εδράζεται αυτή η νέα στρατηγική. Φυσικά προσβλέπουμε όλοι σε αυτή. Επίση, θεωρώ ότι και τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι πολύ πιο ανοιχτά, ιδίω σε ό,τι αφορά τι ανάγκε και τι απαιτήσει τη οικονομία. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία Επομένως ελπίζω η δεκαετία, η δεύτερη της μεταρρύθμισης να είναι πιο πολύ εστιασμένη στον εξυγχρονισμό και την επικαιροποίηση της διδακτέας ύλη σε ό,τι αφορά την ουσία και όχι μόνο να είναι μια τεχνική εναρμόνιση. Εν κατακλείδη, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στον περαιτέρω εξυγχρονισμό της ανώτερης εκπαίδευσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, πρώτα απ' όλα σα ευχαριστώ για την διαθεσιμότητά σα απέναντί μα, πράγμα το οποίο μα επιτρέπει να εργαστούμε σε ένα καλύτερο πλαίσιο. Θα σταθώ σε δύο σημεία από αυτά που αναφέρατε προηγουμένως. Όσον αφορά την εκπαίδευση για τα πανεπιστήμια, έχουμε την αίσθηση ότι ο 21ος αιώνα στην Ευρώπη άρχισε με πολλές αδυναμίες για τα πανεπιστήμια που δεν κατάφεραν να προσελκύσουν τους καλύτερους ερευνητές, τους καλύτερους φοιτητές και το καλύτερο ε, πνευματικό δυναμικό, όχι μόνο της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη χάνουν φυσικά φοιτητές που πάνε αλλού, που ίσως είναι και φυσιολογικό, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε λιματικοί σε αυτό το ισοζύγιο, αλλά δεν, καταφέρνει, ε, δεν καταφέρνουμε να ε, προσελκύσουμε ερευνητές στα πανεπιστήμια μας από άλλα μπλοκ και αναφέρομαι ιδιαίτερα στην Ασία και στην Νότια Αμερική. Και ήθελα λοιπόν να ε, σας ρωτήσω πώς θα κάνετε αυτή την απογραφή στην οποία αναφερθήκατε. Με βάση ποια κριτήρια θα κρίνετε τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία των πανεπιστημίων μας, όπως είπατε. Και όσον αφορά τις υποτροφίες, σε βάση ποια κριτήρια θα πρέπει να προτείνουμε να δίνονται. Τώρα, για τους ε, δημιουργικούς κλάδους, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι είναι απολύτως σημαντικό να χαραχτεί ένα, δημο... ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ε, πολλές... Ε, πολλά πράγματα έχουν γίνει αλλά δεν έχουμε προωθήσει ε, πραγματικά τη δημιουργικότητα. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας ε, ε, κυρία Επίτροπε ότι η αγορά δεν αρκεί και ότι ε, πρέπει το δημόσιο, ο δημόσιος τομέας να κάνει κάτι για τις νέες επενδύσεις, ιδίως για τον ψηφιακό τομέα. Uh, ο κ. Παπενικολάου, τελευταίος σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, πράγματι είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας για μας εδώ και η ενημέρωση την, ε, την οποία μας παρέχεται για την περαιτέρω πορεία και, την, και το σχεδιασμό της δικής σας Επιτροπής. Θα ήθελα να αναφερθώ σε εκείνα τα παιδιά που εγκαταλείπουν προώρα το σχολείο. Ένα πολύ σημαντικό και μείζον ζήτημα, παρότι ζούμε σε σύγχρονες κοινωνίες, δυστυχώς τα νούμερα είναι αποθαρρυντικά. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι στο προϋπολογισμό που ψηφίσαμε δεν υπάρχει κάποια γραμμή του προϋπολογισμού για το θέμα αυτό ε, και δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Το δεύτερο αφορά, από τη μία έχουμε την πρόληψη του φαινομένου, από την άλλη έχουμε την αντιμετώπιση του προβλήματος για εκείνα τα παιδιά που διαπιστώνεται ότι έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Ε, προγραμματίζει η Επιτροπή κάποιο σχεδιασμό και την ανάλυση πρωτοβουλειών για εκείνο που οι κοινωνιολόγοι αποκαλούν κοινωνική χαρτογράφηση για τα παιδιά δηλαδή που έχουν φύγει από το σχολείο να δούμε πού πάνε μετά. Καταλήγουν στο περιθώριο και σε διάφορες δραστηριότητες που όλοι καταλαβαίνουμε ποιες είναι. Η τεχνική κατάρτιση που μπορεί να τους προσφερθεί από τα κράτη-μέλη είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Σχεδιάζει η Επιτροπή κάτι από αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ich Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ε, θέλω και εγώ να ρωτήσω κάτι. Αναφερθήκατε σε υποτροφίες ευρωπαϊκές που θέλετε να εισαγάγετε. Μα έχουμε ευρωπαϊκές ε, υποτροφίες στο πρόγραμμα Erasmus Mundus. Μικρές είναι αυτές, αλλά εντάξει, υπάρχουν. Τώρα αυτές οι υποτροφίες οι οποίε αναφερθήκατε εσεί, πότε θα δίνονται, πώς και σε ποιον, μέσα στα πλαίσια ποιου προγράμματος ή εκτός προγράμματος. Αυτό που μου φαίνεται καλό είναι ότι επί τη ευκαιρία αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Καλό, αυτοί έχουν λεφτά, εμείς δεν έχουμε. Τι έχετε λοιπόν κατά νου εσείς. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα ερωτήματα. Εύστοχα. Ας ξεκινήσω με την Ανατολική Εταιρική Σχέση. Το πρόγραμμα το πολιτιστικό δρομολογήθηκε το 2010. Το πρώτο τμήμα επικεντρώνεται στην παροχή τεχνικής βοήθειας, περιφερειακή παρακολούθηση, μονάδα υποστήριξης. Το δεύτερο τμήμα είναι προκήρυξη διαγωνισμού για την ενίσχυση των δυνατοτήτων ε, στον πολιτιστικό τομέα. Στο πλαίσιο της ανατολικής δράσης για το 2010 του EMP. 12 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προπολογισμό. Αυτά είναι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Χθε ήμουν στο Τωρίνο, συμμετείχα σε μια συνάντηση με το ETF και τους εταίρους μας, τους εκπροσώπους ε, της γειτονίας από την ε, παιδεία και τον πολιτισμό. Συζητήσαμε μαζί τους μεταξύ άλλων τους τρόπους ε, με τους οποίους θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε όσον αφορά την πτυχή της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Από τη δική μας πλευρά η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης Ιδίω ε, μετά την ολοκλήρωση τη ε, της εκπαίδευση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, λοιπόν, ε, πρόκειται για μια εταιρική σχέση που η συνεργασία μας πηγαίνει πολύ καλά. Α έλθω στον αθλητισμό. Το θέμα του αθλητισμού πρέπει να σας πω ότι δεν είναι τόσο σοφερά τα πράγματα. Όταν συμπεριλήφθη ο αθλητισμός στη συνθήκη της Λισαβόνας, Χωρήθηκε μένει αρμοδιότητα σε εμά, όχι όμω και ο προπολογισμό που θα μπορούσαμε να διαθέσουμε για τον αθλητισμό. Για το εναπομένων λοιπόν μέρο ε, του τρέχοντο πλαισίου δεν έχουμε χρήματα για τον αθλητισμό μέχρι το 2013. Ίσως όμως τελικά να είναι και καλύτερα τα πράγματα. Γιατί. Γιατί έχουμε τις παρασκευαστικές ενέργειες οι οποίες ε, συνεχίζονται και όπως είπα θα συνεχιστούν μέχρι το 2012. Κατόπιν θα έχουμε την αξιολόγηση επιπτώσεων, η οποία θα βασίζεται στα στοιχεία τα οποία θα έχουμε συγκεντρώσει από τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και η ανακοίνωση ουσιαστικά θα ανοίξει το δρόμο για το πρόγραμμα το ειδικό για τον αθλητισμό υπό τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές. Επομένως ευελπιστώ ότι με την ανακοίνωση που ελπίζω να εγκρίνουμε στις αρχές Δεκεμβρίου και με τις προπαρασκευαστικές ενέργειες θα μπορούμε να στοχεύουμε σε ένα ουσιαστικό πρόγραμμα για τον αθλητισμό μετά το 2013. Σε ό,τι αφορά την ανώτερη εκπαίδευση. Είσατε για την ανώτατη εκπαίδευση και κατά πόσον έχουμε κάποια ε, υπόψη μας για να δώσουμε έμφαση στα, στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδέ. Πρέπει να τονίσω και πάλι ότι εδώ είναι τα κράτη-μέλη που αποφασίζουν και τα, φυσικά τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τι σπουδέ θα επιδιώξουν. Όμω πιστεύω ότι με το νέο mapping, όπω λέμε, των πανεπιστημίων, διότι όπως είναι σήμερα τα πανεπιστήμια, είναι οργανωμένα όλα μαζί. Δεν ξεχωρίζουν μεταξύ πανεπιστημίων, τα οποία είναι ακαδημαϊκά ιδρύματα ή πανεπιστήμια με επαγγελματική εκπαίδευση ή τεχνικά πανεπιστήμια ή πανεπιστήμια τα οποία δίδουν έμφαση στις ανθρωπιστικές σπουδές. Τώρα, με αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε και αυτή τη στιγμή διεξάγουμε μία μελέτη, πολύ μεγάλη μελέτη, η οποία πιστεύουμε θα είναι έτοιμη μέχρι τον Μάιο του 2011 και βάσει αυτής της μελέτης θέλουμε να ξεχωρίσουμε τα πανεπιστήμια σε κατηγορίες ανάλογα με τον προσανατολισμό των πανεπιστημίων. Και εκεί φυσικά και η αναγνώριση των ε, πανεπιστημίων θα γίνεται από την ίδια ε, ε, από την ε, ίδια κατηγορία πανεπιστημίων. Δεν θα συγκρίνουμε δηλαδή πανεπιστήμια τεχνικά με εκείνα που είναι ανθρωπιστικών σπουδών, αλλά τη ίδια κατηγορία. Αυτό πιστεύω από μόνο του θα βοηθήσει στο να δοθεί έμφαση στα, και στι κοινωνικέ και ανθρωπιστικέ σπουδέ. Μου θέσατε και ένα ερώτημα σχετικά με τον εξυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης. Είπατε, δεν θυμάμαι ποιος το είπε ακριβώς, ότι χάσαμε χρόνο. Εγώ δεν θα το έλεγα. Γιατί η διαδικασία της ε, Μπολόνια χρειαζόταν το χρόνο αυτό. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν χώρες, υπάρχουν πανεπιστήμια, τα οποία δεν έχουν καταφέρει να εξυγχρονίσουν τα πανεπιστήμια τους με βάση τη διαδικασία της Μπολόνια. Τώρα όμως δίνουμε έμφαση στον εξυγχρονισμό της διδακτέας ύλη, στη διακυβέρνηση, στην αυτονομία, στη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Αυτό εννοούμε όταν μιλάμε για εξυγχρονισμό του πανεπιστημίου. Θέλουμε επίσης τα πανεπιστήμια να αποκτήσουν ένα πιο διεθνή χαρακτήρα, να μπορούν να ανταγωνίζονται στη διεθνή σκηνή. Και νομίζω ότι είναι κάτι πραγματικά αναγκαίο. Τώρα πολιτιστικός και δημιουργικός κλάδος. Όπως γνωρίζετε, ολοκληρώσαμε την ανοιχτή διαβούλευση. Είχαμε ένα πολύ καλό ποσοστό ανταπόκρισης και τώρα αναλύουμε τα στοιχεία τα οποία συλλέξαμε με την ανοιχτή αυτή διαβούλευση. Και πρόκειται να εκπονήσουμε ένα βασικό έγγραφο εργασίας βάσει του οποίου θα αποφασίσουμε ποιες δράσεις, ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναλάβουμε ούτω ώστε να βοηθήσουμε και να προωθήσουμε τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό κλάδο. Σε σχέση με το θέμα αυτό, συνεργάζομαι και τον Επίτροπο Χάν για να δούμε πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κονδύλια. Πώς θα μπορούσαν επίσης τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα περιφερειακά κονδύλια για τον τομέα του πολιτισμού. Γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν στη διάθεσή τους ε, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Τώρα έρχομαι στο ερώτημα της ε, πρόορης εγκατάλειψης ε, του σχολείου. σχολείο νωρίς είναι κυρίως παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση για πολλούς και διάφορους λόγους. Ε, οι μελέτες μας δείχνουν ότι δεν είναι ένας ο λόγος, αλλά διάφοροι λόγοι. Άλλοι διότι οι, δεν έχουν την ενθάρρυνση που χρειάζονται από, το, από την οικογένεια και το σπίτι. Άλλοι διότι δεν βρίσκουν το σχολείο αρκετά ενδιαφέρον για να τους κρατήσει στο σχολείο και για διάφορους λόγους. Αυτό που θα κάνουμε του χρόνου είναι θα κάνουμε μία ε, πρόταση προς τις ε, χώρες μέλη που να τους δίδουμε διάφορες ιδέες το πώς να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο διότι δεν έχουμε μία συνταγή η οποία να αντιμετωπίζει όλες τις περιπτώσεις. Είναι, όπως είπα, ανάλογα με τον περιπτώσιο Και εφόσον θα δώσουμε στις χώρες μέλη διάφορες ιδέες, οι χώρες μέλη θα ε, επιλέξουν εκείνες τις συνταγές που είναι οι πιο κατάλληλες για την περίπτωση που έχουν να αντιμετωπίσουν. Ε, επίσης για τα παιδιά τα οποία εγκαταλείπουν το σχολείο θα τους δώσουμε και μία ε, πρόταση για το πώς θα επαναφέρουν αυτά τα παιδιά στην εκπαίδευση. Διότι ορισμένα εγκαταλείπουν τελείως την εκπαίδευση, αλλά όμως είναι παιδιά τα οποία έχουν ε, ύφεση για μάθηση, αλλά χρειάζονται ε, διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Ε, και γι' αυτό νομίζω το να κάνουμε το σχολείο πιο, ε, αν θέλετε, ενδιαφέρον για αυτά τα παιδιά. Ένα παράδειγμα να σας πω. Σχολεία τα οποία δίδουν έφαση στον αθλητισμό. Για πάρα πολλά παιδιά τα οποία εγκαταλείπουν το σχολείο, αυτόν και από μόνον του είναι τρόπος να τα κρατήσει στο σχολείο. Και δεν σας το λέγω διότι εγώ το ξέρω, αλλά οι μελέτες το έχουν αποδείξει αυτό. Γι' αυτό και έχουν διάφορα κοινωνικά προγράμματα το πώς να χρησιμοποιήσουν τον αθλητισμό και άλλα μέσα, τις τέχνες, ε, για να κρατήσουν τα παιδιά ή να επαναφέρουν τα παιδιά στην μόρφωση. Ε, αυτό που είπα, Doris, για την ενίσχυση προς τους φοιτητές δεν είναι υποτροφίες, είναι δάνεια στους φοιτητέ για να αναπτύξουν μια κινητικότητα. Το συστάμε το θέμα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους από εκεί και επίσης από τοπικές και εθνικές ε, τράπεζες για να προσφέρουμε δάνεια σε φοιτητές που θέλουν να κινηθούν, να μετακινηθούν, αλλά δεν έχουν τα χρήματα που χρειάζεται ή για τους οποίους τα χρήματα που δίνουμε εμείς από τα διάφορα προγράμματα δεν αρκούν για να πάνε στη χώρα στην οποία θέλουν να πάρουν. Χρειάζεται λοιπόν μια επιπλέον ενίσχυση των φοιτητών αυτών. Και βέβαια όταν ολοκληρώσουμε το σχέδιο θα σας το υποβάλουμε και μπορούμε να το συζητήσουμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει πρόεδρο. Δέκα συναδέλφους έχω καταγράψει. Όχι, δεν ήσασταν εδώ, δεν μπορείτε να υποβάλλετε ερώτηση. Τώρα να, να έρθετε δηλαδή μόλις, να, μόλις έρθετε να βάλετε και ερώτηση όχι. Δέκα. Και σας παρακαλώ, αυτά που έχουν ερωτηθεί μην τα ξαναρωτήσετε. Ο κύριος Μπόρης. Ε, e, ε, Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το τόσο φιλόδοξο αυτό ε, πρόγραμμα. Το πρώτο σημαντικό θέμα, η Ευρώπη του 2020. Εσείς αναφερθήκατε ε, μια εν ώψη της ε, διαδικασίας Πολώνια και των αυξανόμενων ανταγωνισμών μεταξύ των διεθνών πανεπιστημίων ιδίω ανταγωνισμό με την Αμερική και την Ινδία και την Κίνα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα δεν είναι η ποιότητα, αλλά η ποσότητα, γιατί ο στόχος ήταν να θα αυξήσουμε τον αριθμό των παιδιών που είναι στα σχολεία κατά 10%. Εσείς τι πιστεύετε, ε, μπορούν τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα για να το πετύχουν αυτό μέσα σε 10 χρόνια. Δεν είναι και τόσο πολλά τα 10 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι υπερβολικά αισιόδοξο. Γιατί ε, αυτός ο χρόνος θα μας χρειαστεί για να έχουμε τους δείκτες από την Αμερική. Και δεν μιλάω για αυτούς από την Κίνα. Εμείς θέλουμε να μειώσουμε το κοινωνικό ε, ε, αποκλεισμό με τον εισαχθούν όλοι στο ψυχιακό κόσμο. Μπορούμε έτσι να πετύχουμε ακόμα και μικρούς, ε, μικρούς στόχους. Εσείς έχετε κατά νου, παραδείγματος χάρη, να χρησιμοποιούνται μια συνοχή για τον κινηματογράφο. Ευχαριστώ. Η κυρία Καμερέβερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Μία παράκληση και μία ερώτηση. Η παράκληση αφορά την ένταξη της πολιτιστικής πολυμορφίας ή γενικά των πολιτιστικών πτυχών στο σύνολο της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι που σας απασχολεί ιδιαίτερα και είναι απόλυτα σαφές και στο δικό σας τομέα εργασίας ότι πραγματικά ε, είσαστε υπέρμαχος ε, του πολιτισμού και των πολιτιστικών θεμάτων. Δυστυχώς βλέπουμε ότι όταν πρόκειται για τομεί οι οποίοι δεν άπτονται άμεσα του πολιτισμού, το θέμα το πολιτιστικό παραβλέπεται. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να επιδράσετε κατά το δυνατόν ε, πάνω στους επιτρόπους συναδέλφους σας ούτως ώστε το θέμα της πολιτιστικής πολυμορφίας να λαμβάνεται υπόψη σε όλους τους τομείς πολιτικής Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορεί να μην χρειάζεται κάθε φορά εμεί να παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη. Το δεύτερο αφορά τον αθλητισμό και έχω μια ερώτηση σχετικά με κάτι που εξετάσαμε ενημερισμένη συνεδρίαση γιατί εξετάσαμε μια μελέτη συνδίκηση της Αβώνας και αθλητισμός που νομίζω μας απογοήτευσε όλους γιατί διευκρινίστηκε απόλυτα ότι τουλάχιστον μέσα στα πλαίσια της μελέτης αυτής δεν θεωρήθηκε ότι είναι αναγκαίο να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο νομοθετικό τομέα για τον αθλητισμό. Στο Κοινοβούλιο, παραδείγματο χάρη, εμεί γκρίναμε μια παράκληση προς την Κομισιόν να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ε, χωρίχης αδείας σε εκείνους που ο, ασχολούνται με την ε, μεταβίβαση και τη μεταφορά των αθλητισμών από μια χώρα στην άλλη. Ε, αυτό είναι πάρα σημαντικό ιδίως για τους νέους αθλητές ε, και ξέρουμε ότι ε, σε πολλές χώρες οι διάφορες αθλητικές οργανώσεις αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν. Και αυτό που είδαμε μέχρι στιγμής δεν αρκεί, γιατί ίσως μεγάλες οργανώσεις μπορούν να αυτό διοργανωθούν, αλλά υπάρχουν και μικρές οργανώσεις που δεν έχουν τον απαραίτητο μηχανισμό και ελπίζουν ότι εμείς θα βρούμε μια λύση. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω ακριβώς σε αυτό το τομέα να δράσει τον του δυνατόν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Μάτουλα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, ήθελα να κάνω μία ερώτηση σχετικά με τη σύνδεση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην εκπαίδευση και στον αθλητισμό στο σχολείο. Το σχόλιο μου βασίζεται σε μια απλή διαπίστωση. Πριν από χρόνια, ο αθλητισμός ε, τα σπορ τραβούσαν τα παιδιά προς το σχολείο. Σήμερα φαίνεται ότι οι πρακτικές του αθλητισμού φοβίζουν ένα μεγάλο ρυθμό παιδιών και εξού και ένα φαινόμενο πολύ ε, σοβαρό που το αναφέρετε που είναι η εγκατάλειψη του σχολείου και ένα άλλο πολύ εξίσου σοβαρό φαινόμενο που είναι η παχυσαρκία μεταξύ των ε, νεότερων παιδιών. Πιστεύω λοιπόν ότι ο αθλητισμός μπορεί και να τραβήξει τα παιδιά στο σχολείο του νέου στο σχολείο και να αντιμετωπιστεί έτσι και το άλλο πρόβλημα. Γι' αυτό ήθελα να σα ρωτήσω ποιος, ε, ποια είναι η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική σα σχετικά με τη σύνδεση ανάμεσα στο σχολείο και στον αθλητισμό και ποιο είναι ο ιδανικό αριθμό ορών, παραδείγματο χάρη στο σχολικό πρόγραμμα αθλητισμού. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Με κάθε σεβασμό ε, μάλλον από σεβασμό προς αυτά που είπατε, ε, θα επικεντρωθώ μόνο σε δύο σημεία, παρόλο που είχα περισσότερα. Αναφέρθηκε η Επίτροπος σε ένα σύστημα χαρτογράφησης των ισχυρών και σημείων και των αδυναμιών των πανεπιστημίων. Αυτό χρειάζεται πάρα πολύ σήμερα, γιατί πολύ συχνά τα πανεπιστήμια στις χώρες μας ε, ζουν ε, σε απομόνωση και δεν αποδίδουν όπως θα έπρεπε. Ένα νέο σύστημα ταξινόμηση, αξιολόγηση των πανεπιστήμιων ε, χρειάζεται. Παρόλο που πολλά πανεπιστήμια δεν προσαρμόζονται όπως θα έπρεπε. Στο Σαντιέγκο πριν από μερικούς ε, μήνες ε, συζητήθηκε για το θέμα ε, της διασύνδεσης ανάμεσα στα πανεπιστήμια και στον επιχειρηματικό κόσμο. Για κάτι τέτοιο θα έπρεπε να το ενθαρρύνουμε. Δεύτερον, για τη διαβίου μάθηση και την ε, κοινωνία που θα βασίζεται στη μάθηση με συμμετοχή όλων ε, θα, με ενδιαφέρει περισσότερο να ακούσω κάτι σχετικά με αυτό. Και τρίτον, αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι για τον αθλητισμό. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να είναι ότι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών θα έπρεπε να ε, έχουν κάποιο είδους ε, σωματική άσκηση. Ε, μέχρι το 2020. Αυτό δεν σημαίνει επαγγελματικό αθλητισμό. Έστω και αν ε, ε, λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα σκάνδαλα και τα, τις υπέρογες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο το θέμα είναι πώς μπορούμε να έχουμε περισσότερους ανθρώπους να ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που λέτε ότι θα είναι ε, το φλάξι αυτό για σας, η εμβληματική σας δράση. Ο κύριος Στογιάννοφ, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση. Ε, χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Εκτελεστικής Επιτροπής στον τομέα της ε, εκπαίδευση και του πολιτισμού. Χαίρομαι για τις πρωτοβουλίε αυτές. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Η, η ζωή των ανθρώπων σήμερα εξαρτάται όσο πάει και περισσότερο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει κάποια πρωτοβουλία στον τομέα αυτό συγκεκριμένα δηλαδή στην αναζήτηση σημείων επαφής μεταξύ πολιτισμού και ΜΜΕ. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε εδώ κάποια μεταρρύθμιση στα πλαίσια τις οποίες όχι μόνο οι πολίτες αλλά και οι πολιτικές αυτές θα μπορούσαν να προωθηθούν τα σημεία αυτά επαφής. Εγώ θα μπορούσα να παραιτηθώ από την ερώτησή μου γιατί είχα μια ερώτηση για τον αθλητισμό και νομίζω ότι η Επίτροπος έχει καταλάβει πόσο μας απασχολεί αυτό το θέμα. έκανε και οι συνάδελφοι ε, τις σχετικές ερωτήσεις. Ε, επομένως δεν επιμένω στην ερώτησή μου. Ευχαριστώ για την Επίτροπο για αυτά που μας είπε. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Ε, συνδέομαι με την ε, παρατήρηση της κυρίας ε, Παλιατέλη σχετικά με τις ανθρωπιστικές σπουδέ ε, ε, στα πλαίσια της ε, ανώτερης εκπαίδευσης και της πανεπιστημιακής πιο συγκεκριμένα. Μία ερώτηση κυρία Επίτροπε. Σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή εργαζόμαστε για θέματα που αφορούν τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Παραδείγματο χάρη το European Heritage Label. Στη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει κάποιο μηχανισμό για να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα ε, στους δύο αρμόδιους επιτρόπους, δηλαδή πολιτισμού και τουρισμού. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επίτροπο για αυτά που είπε για τον εξυγχρονισμό των πανεπιστημίων. Ήθελα να σας αναφέρω μια ανησυχία μου. Πιστεύω ότι η διαδικασία της Μπολόνια προχωράει πάρα πολύ αργά και ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης δεν κάνουν αρκετά πράγματα. Τα πανεπιστήμια αισθάνονται μόνα τους στο, στη Βόρεια Ευρώπη, στην Κεντρική Ευρώπη, τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Και εδώ και εκεί σε άλλα σημεία ε, της ε, Ευρώπης υπάρχουν κάποια θετικά σημεία, αλλά υπάρχει ένα μέρος της Ευρώπης που δεν πιστεύει στη διαδικασία της Μπολόνια. Θα σας πω το εξή: Πανεπιστήμια που δεν δίνουν ευρωπαϊκούς τίτλους σπουδών και που δεν εξασφαλίζουν την ε, χρήση αυτών των τίτλων σπουδών στους φοιτητές τους. αυτά τα πανεπιστήμια δεν πρέπει να βοηθούνται γιατί αρνούνται τον βασικότερο ρόλο τους. Γιατί είναι κολλημένα τα πανεπιστήμια αυτά σε μια ξεπεραμένη σε μια ξεπερασμένη ιδέα για το ρόλο τους. Δηλαδή, ε, θα πρέπει να δοθούν κινητρά σε όλους αυτούς που δίνουν τίτλους ήδη, χωρίς να παίρνουν καμία ενίσχυση. Δεύτερον, quality assessment. Διότι και η χαρτογράφηση αυτή θα βοηθήσει πάρα πολύ για να δούμε ποια είναι τα πανεπιστήμια που δίνουν τίτλους που δεν έχουν ισχύ παρά μόνο μέσα στο εσωτερικό της χώρας τους και τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε επίτρεπε, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα ε, που θίξετε στου τομεί ε, πολιτισμού και δημιουργικότητα, γιατί η Κομισιόν μα πρότεινε κάποια πρωτοβουλία. Η πράσινη βίβλο οδήγησε σε αντιδράσει έντονε, πραγματικέ διαβουλεύσει και βλέπουμε πόσο διαφορετικές είναι οι βιομηχανίες αυτές οι τομείς και στο μέγεθός και όσον αφορά το ρόλο τους που παίζουν στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Πώς θα λάβουμε υπόψη μας αυτές τις τόσο μεγάλες διαφορές. Είναι ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό που θα πρέπει να απαντήσουμε με τη στρατηγική που θα εγκαθιδρύσουμε για να συνοδεύσουμε τις βιομηχανίες αυτές. Κατόπιν θα ήθελα να υποστηρίξω την ε, παρέμβαση του συναδέλφου Ζωμαρή Καβαντά όσον αφορά την απαραίτητη εταιρική σχέση που θα πρέπει να υπάρχει με τα κράτη-μέλη και την τοπική αυτοδιοίκηση που θα μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε τους τομείς ε, δημιουργικότητας και πολιτισμού, ιδίως όσον αφορά το θέμα της δημιουργικότητας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, κάτι πάρα πολύ χρήσιμο που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι η κινητικότητα. Στις βιομηχανίες αυτές αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς μπορούμε να θερύνουμε την κινητικότητα αυτή προστατεύοντας την, ε, προωθώντας συγγνώμη, την προστασία της δημιουργίας. Και θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει δυνατότητα με τον Επίτροπο Φανεσάν μέσα στα πλαίσια των ε, μέιο Συνοχής ε, να εκμεταλλευτούμε κάποιες δυνατότητες για να υποστηρίξουμε την πολιτιστική βιομηχανία. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ο κύριος Φυσάς. Εκτός μικροφώνου. Έλεγα λοιπόν, ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή τα αεροπλάνα δεν κυκλοφορούν πολύ καλά. Ήθελα να σχολιάσω κάτι, δεν ξέρω αν υπόθηκε προηγουμένω. Πρόκειται για το copyright, τα δικαιώματα πνευματική διοκτησίας. Ξέρετε ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αφορά διάφορους τομείς, νομικές υπηρεσίες, βιομηχανία, αλλά και στον πολιτισμό. Πρέπει να βρούμε και εμείς πώς θα μπορούσαμε την σωστή αμοιβή που θα πρέπει να έχουν οι δημιουργοί να τη συνδυάσουμε με την ελευθερία πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παραδείγματο χάρη τώρα στην Ισπανία Είχαμε ένα ψηφιακό τέλος, το οποίο πρόσφατα ε, κυρώθηκε ως ρύθμιση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις. Ε, δηλαδή θεωρήθηκε παράνομο το τέλος αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η δική σας θέση απέναντι σε αυτά τα γεγονότα και πώς ε, προχωρούν οι συνεδριάσεις μεταξύ των διαφόρων επιτρόπων που είναι αρμόδιοι για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Για εμάς μάλιστα είναι ένα θέμα που στην Επιτροπή Πολιτισμού μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του δημιουργού. Είναι σαφέ ότι ο κ. Μπαρνιέ είναι υπεύθυνο για το τομέα αυτό. Ελπίζω όμω ότι η Επίτροπο μας ε, έχει πάντα κατά τον τομέα του πολιτισμού. Η κυρία Κώστα. Ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο κύριε Βασιλείου γιατί εστίασε σε τρία θέματα που είναι πραγματικά στρατηγικά. Πιστεύω ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια φάση πάρα πολύ σημαντική γιατί θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο όλη αυτή την ε, πολιτική της, ε, του πολιτισμού και της ε, εκπαίδευσης μέσα στη στρατηγική του 2020. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν που αναφέρατε για μένα είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι πρέπει να ξαναδρομολογήσουμε αυτές τις πολιτικές γιατί αφορούν τομείς που είναι είναι για μας η πιο στρατηγική. Ε, και τα λέω αυτά γιατί εδώ στην Επιτροπή μας, ε, ε, στην η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον, συμμερίζεται την άποψή μας αυτή. Για την νεολαία σε κίνηση ήθελα να πω ότι μιλάμε για τον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης και πολιτισμού. Το Youth on the Move πρέπει να είναι μια απάντηση στο θέμα αριστεία και ισότητα, όπως είπατε, και στο δικαίωμα που έχουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά στην κινητικότητα και στην διαβίου μάθηση. Πιστεύω όμως ότι χάρη και στην ε, Επιτροπή, ε, ε, αν είχαμε κάποια ε, κονδύλια περισσότερο για το Youth on the Move ε, από ό,τι για το Erasmus, ε, πάλι είμαστε μακριά από το να δώσουμε ε, τις δυνατότητες που πρέπει να έχουν οι νέοι στην Ευρώπη για την κινητικότητα. Αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα επειδή σαν πηγή και άλλων πόρων πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε και μια ποσοτική ένδειξη πιο ισχυρή για τα ταμεία συνοχής όπως είπε ο προηγούμενο συνάδελφος και πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για ευρωπαϊκές υποτροφίες εργασίας και υποτροφίες σπουδών μέσω του κοινωνικού ταμείου. Ε, πρέπει να σας πω ότι είμαι σχιώδης ηγετρία για, τις, ε, για τους ε, πολιστικούς και δημιουργικούς τομείς και έκανα μια πολύ μεγάλη διαβούλευση και πρέπει να σας πω καταρχάς ότι πολλοί ε, δεν ξέρουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται, δεν παίρνουν τις πληροφορίες και τη σωστή ενημέρωση. Ένα πράγμα όμως είναι σαφές, ότι είναι πάρα πολύ θετικό να το πει αυτό η Ευρώπη καθαρά, ε, να, να μιλήσουμε δηλαδή για τον δημόσιο ρόλο για τις πολιτιστικές και ε, δημιουργικές βιομηχανίες ε, και να μην το αφήσουμε αυτό μόνο στην αγορά. Δεύτερον, το θέμα της αμοιβή ε, του έργου τέχνης, το στάτους του καλλιτέχνη και του δημιουργού που στις 12 από τις 27 χώρες αναγνωρίζεται και ίσως καλό θα ήταν η Ευρώπη να δώσει μια τέτοια ε, κατεύθυνση, το θέμα της ψηφιοποίησης των αιθουσών των κινηματογραφικών και επίσης το θέμα ε, Τη δημιουργικότητα και πάλι. Τώρα, για τον πολιτιστικό τουρισμό, χαίρομαι πάρα πολύ που εγκρίθηκε η προπαρασκευτική μας ε, δράση και πιστεύω ότι η μορφή αυτού του τουρισμού θα προωθήσει τα, τις πολιτικές διαδρομές στην Ευρώπη, θα συμβάλλει στις πολιτικές διαδρομές που πιστεύω ότι είναι, ε, ε, έχει να κάνει με την κληρονομιά κλπ. Πιστεύω ότι το τομέας αυτός πρέπει να βρει χώρο μέσα στους... Ε, δημιουργικούς τομείς. Γιατί ο τουρισμός και η μόδα ε, δεν αφορούν μόνο τη δημιουργικότητα. Και για τον ε, πολιτικό τουρισμό, επειδή στις 27 Σεπτεμβρίου είχαμε την Ευρωπαϊκή ημέρα τουρισμού και επειδή ε, και ο, ο κύριος Ταγιάννη ασχολήθηκε με αυτό το θέμα θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συνεργάζεστε στενά για να υπάρχει πιο μεγάλη συνέργεια ανάμεσα στον πολισμό και τον τουρισμό και, τις, και τους σχετικούς ε, κλάδους, τους οικονομικούς ούτως ώστε το σχέδιο αυτό να γίνει κάτι το πολύ πιο στρατηγικό πράγμα το, με το οποίο συμφωνώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ μια ερώτηση που την σκέφτηκα την ώρα που απαντούσατε προηγουμένως κύριε Επίτροπε όσον αφαιρθεί την κατηγοριοποίηση αυτό τον χάρτη αν θέλετε τη χαρτογράφηση των πανεπιστημίων αυτό κάπως με ενοχλεί. Τι θα πει αυτό. Είναι ταξινόμηση ανα, σύμφωνα με την ποιότητα. Θα υπάρχει μια πύλη αν θέλετε που θα απαριθμεί όλα αυτά που βρίσκει Κάτε ή θα κάνετε και αξιολόγηση αυτόν καλύτερο, αυτόν χειρότερο. Γιατί νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν το θέλαμε. Αν έχετε μια απαρίθμηση όλων των δυνατοτήτων, αυτό μου φαίνεται καλό. Αλλά όχι ανακατηγορία ή ταξινόμηση ή σύμφωνα με την ποιότητα. Αυτό δεν θα μας άρεσε. Τώρα, υποβάλαμε όλες τις ερωτήσεις μας. Σας παρακαλώ να απαντήσετε, Αντρούλα. <laughs> Πολλές ερωτήσεις, ε, να δούμε αν θα μπορέσω να τις απαντήσω. Αν θυμάμαι ό,τι με, ό,τι με ρωτήσατε όλοι. Καταρχάς να διορθώσω κάτι. Δεν πρόκειται για αναθεώρηση της διαδικασίας της Μπολόνια, αλλά για συνέχιση της διαδικασίας αυτής. Σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια, ήμουν ε, στην ετήσια συνδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστήμιου στο Παλέρμο πρόσφατα. Και πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ πολύ άσχολη. Όλοι θέλουν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία της Μπολόνια. Να καταστήσω σαφές το εξή. Η διαδικασία της Μπολόνια είναι διακυβερνητική, δεν είναι μια ενωσιακή διαδικασία. Φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει και προσπαθεί να βοηθήσει τη διαδικασία της Μπολόνια, αλλά δεν είναι δική μα πρωτοβουλία. Όπω και να έχει όμω, τα πανεπιστήμια τώρα, όπω σα είπα, προσπαθούν να εξυγχρονίσουν το πρόγραμμα σπουδών του, τον τρόπο χρηματοδότηση, τη διακυβέρνηση, διαχείρισή του, αν θέλετε και την ποιότητα. Η ποιότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση είναι το ίδιο σημαντική με την ποσοτική, γιατί φυσικά και θέλουμε να ανοίξουμε τα πανεπιστήμια μας σε το δυνατόν περισσότερους φοιτητές. Η ποιότητα όμως για εμά είναι και παραμένει υπαριθμών ένα προτεραιότητα. Τώρα, Δεν θα απαντήσω με τη σειρά των ερωτήσεων, γιατί κάποια ερωτήματα σχετίζονται μεταξύ τους. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα πανεπιστήμια, αφού είμαστε σε αυτό το θέμα, νομίζω κύριε Μπόρις εσείς ήσασταν αυτός που με ρώτησε για την δυνατότητα επίτευξης αυτού του 40% του στόχου αυτού. Ακούστε. Να σας εξηγήσω πώς εμείς εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Κάθε κράτος μέλος διαφέρει. Κάποια κράτη-μέλη προς το παρόν έχουν 15-20% ή κάποιο ισοδύναμο σε ό,τι αφορά τους ε, αποφύτους. Κάποιοι έχουν υπερβεί το 40% και φτάνουν στο 50%. Αυτό λοιπόν το οποίο καλούμε τα κράτη-μέλη να κάνουν είναι να υποβάλουν το δικό τους εθνικό στόχο, λαμβάνοντας υπόψη την αφετηρία, το σημείο κίνησης δηλαδή, τις δυνατότητες που έχουν και έτσι να μας καταθέσουν έναν εθνικό στόχο. Από τις 27 χώρες μέλη, ήδη οι 25 μας έχουν παρουσιάσει τον εθνικό του στόχο. Του χρόνου θα μας υποβάλουν μάλιστα εθνικό πρόγραμμα για το πώς ε, προτίθενται να επιτύχουν αυτόν τον εθνικό στόχο. Ελπίζουμε λοιπόν, και εκεί στοχεύουμε, ελπίζουμε να φτάσουμε σε έναν μεσόρο του 40% αφού βέβαια λάβουμε υπόψη όλους τους εθνικούς στόχους που θα έχουμε λάβει. Η διαφορά μεταξύ των στόχων στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της στρατηγικής της Λισαβόνας, μάλλον της στρατηγικής της Λισαβόνας, νομίζω ότι τώρα είναι σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αποφασίσει ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει την ιδιοκτησία, αν μπορώ να το πω έτσι, της στρατηγικής αυτής. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισαν να περιορίσουν τους στόχους μόνο σε πέντε όχι 23 όπως ήταν στο πλαίσιο της συνθήκης Λισαβόνας. Πολιτισμός τώρα. Να σας ευχαριστήσω που αναγνωρίσατε ότι κάνω ό,τι μπορώ για τον τομέα του πολιτισμού. Κατόπιν των δικών μου προσπαθειών, πραγματικά έχουμε συμπεριλάβει πάρα πολύ προσπάθεια, πάρα πολλά στοιχεία στις βασικές ε, πρωτεύουσες πρωτοβουλίες, flagship initiatives όπως τις λέμε. Έχουμε την καινοτομία, την περιλάβαμε, ψηφιακή ατζέντα, νέες δεξιότητες για νέες ε, θέσεις εργασίας που θα υποβάλουμε και επίσης η βιομηχανική πρωτοβουλία του κυρίου Ταγιάννη. Γιατί θέλουμε και εκεί να έχουμε κάτι και για τον πολιτιστικό τουρισμό επίσης. Κάνω ό,τι μπορώ λοιπόν. Μίλησα επίσης με την ε, Βαρόνη Άστον. Σας είπα ότι θέλω να μιλήσω μαζί της για να έχουμε έναν συγκεκριμένο έναν ειδικό τομέα στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης που θα ασχολείται ειδικά με τον πολιτισμό γιατί θέλουμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή εικόνα του πολιτισμού της ε, ποικιλομορφία, της πολυμορφίας σε σχέση με τους εξωτερικούς μας εταίρους. Και φαίνεται ότι η κυρία Άστον ε, είναι ευνοϊκά διακείμενη. Δεν την έχω ακόμη συναντήσει στις ε, Βρυξέλλες, ελπίζω σύντομα να έχω την ευκαιρία. Επίσης, όπως πολύ σωστά είπατε, πάντοτε πρέπει να προσπαθούμε με τους ε, ομολόγους μου επιτρόπους να συμπεριλαμβάνουμε τη διάσταση του πολιτισμού σε όλες τις πολιτικές. Αθλητισμός. Δεν θέλω να σας αποκαλύψω πράγματα που δεν είναι ακόμη οριστικά αλλά μπορώ να σας δώσω μία ένδειξη για το τι θα περιλαμβάνει, ποιες θα είναι οι βασικές ιατρές γραμμές της ανακοίνωσης για τον αθλητισμό. Σίγουρα θα προάγει την κοινωνική και εκπαιδευτική λειτουργία του αθλητισμού. Οι αθλητικές δομές και ειδικότερα αυτές που έχουν να κάνουν με θελοντική δραστηριότητα και με τον απλό πολίτη θα είναι προτεραιότητα. Θα, προωθήσουμε επίσης ε, το fair play, την ανταγωνιστικότητα, την άμυλα στον αθλητισμό ε, την ακαιρεότητα τόσο τη σωματική όσο και την ηθική των αθλητών. Καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης για παράδειγμα, θα είναι μία από τι βασικέ μα δραστηριότητε. Ε, επίσης, θα προωθήσουμε το διάλογο και τη συνεργασία με τους αθλητικούς φορείς. Είναι κάτι που ήδη πράττουμε, αλλά ελπίζουμε σύντομα να συμφωνήσουμε και σε έναν τρόπο που θα μας βοηθήσει να διαρθρώσουμε καλύτερα το διάλογο που έχουμε και με το αθλητικό κίνημα και με τους αθλητικούς φορείς. Για τον κύριο Φίσας. Πράγματι, τα πνευματικά δικαιώματα, το copyright, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για εμάς, για τον πολιτισμό. Και θέλουμε να προστατεύσουμε, θέλουμε να προστατευθούν τα δικαιώματα δημιουργού εν γέννη. Πάντως, πραγματικά, ε, ήταν πολλοί οι επίτροποι που ασχολούνταν. Ο επίτροπος Μπαρνιέ νομίζω ότι θα ξεκινήσει μια ανοιχτή διαβούλευση για το θέμα αυτό πάρα πολύ σύντομα και για όλου, ελπίζουμε, μάλλον ελπίζουμε όλοι να συμμετέχουν σε αυτή τη διαβούλευση γιατί θέλουμε να συμπεριληφθούν και να ληφθούν υπόψη όλε οι πτυχέ. Δεν μπορώ να σα πω ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα τη διαβούλευση. σίγουρα όμω θα ληφθούν υπόψη και τα δικά μα ζητήματα. Γι' αυτό μπορώ να σα διαβεβαιώσω. Θα σας παρακαλέσω όμως να λάβετε και εσείς μέρος στη διαβούλευση αυτή. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε την, την συμβολή όλων όσων ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό. Και μια και μιλάω για τον πολιτισμό, να σας διαβεβαιώσω ότι πολύ σύντομα θα υποβάλουμε μαζί με την ανακοίνωση για τον κινηματογράφο. Προωθούμε βέβαια την ψηφιοποίηση των ε, αιθουσών κινηματογράφου, βοηθώντας μικρούς ε, κινηματογράφους που δείχνουν ευρωπαϊκές ταινίες, να βοηθήσουμε στην ψηφιοποίησή τους. Αλλά θέλουμε και να καταλήξουμε για το Ταμείο Εγγύησης Πίστοσης. Με και Ισπανία προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους κινηματογράφους να παίρνουν ε, κάποιες ε, πιστώσεις, κάποια δάνεια από τις τράπεζες. Σύντομα θα προχωρήσει λοιπόν και αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα το δικό σας ερώτημα, Πντόρης, μιλάμε για χαρτογράφηση των πανεπιστημίων. Αυτό προωθούμε. Όπως είπα, θέλουμε να δώσουμε στους φοιτητές μια πολύ σαφή εικόνα και ιδέα της προσφοράς που υπάρχει ποια πανεπιστήμια προσφέρουν τι και επομένως θέλουμε να έχουμε μια κατάταξη ουσιαστικά των πανεπιστημίων που θα επιτρέπει στους φοιτητές να επιλέγουν με τα γνώσεως. Και όπως ξέρετε διεξάγουμε μια μελέτη η οποία ξεκίνησε ε, επί γαλλικής προδιαστέθη το αίτημα αυτό Ελπίζουμε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Άνοιξη η μελέτη αυτή και βέβαια με βάση τα αποτελέσματά της, νομίζω 120 πανεπιστήμια συμμετέχουν σε αυτήν, θα γνωρίζουμε περισσότερα για την πορεία που θα ακολουθήσουμε στη συνέχεια. Δεν ξέρω ακριβώς αν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια νέα κατάταξη των πανεπιστημίων ή θα είναι μια απλή χαρτογράφηση. Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ πηγαίνουμε προς το να είναι μια χαρτογράφηση και όχι κατάταξη, ταξινόμηση, αξιολόγηση ουσιαστικά. Και η Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε την πλήρη εικόνα τώρα του πολύ δύσκολου έργου σας. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πελινιέρ, er έχει δίκιο. Το θέμα της διαδικασίας Μπολόνια δεν είναι θέμα της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση της Κομισιόν ή του Κοινοβουλίου. Είναι ένα εθνικό πανεπιστημιακό πρόβλημα και αυτή τη στιγμή ούτε η εθνική πολιτική ούτε τα πανεπιστήμια έκαναν ό,τι έπρεπε να έχουν κάνει πρωτού ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Ούτε προσαρμόσανε το διδακτέα ύλη, ούτε βοηθήσαν να υπάρχει καλύτερη διακυβέρνηση των πανεπιστήμιων. Τεράστιο πρόβλημα λοιπόν το διδακτεα ηλί ουτε βοηθησαν τώρα έχουμε μετά από 10 χρόνια μπροστά μα. Εκτό από τι σκανδιναβικέ χώρε έχετε δίκιο κύριε Μπερλίνγκερ, όταν είχα πάει στο Πανεπιστήμιο Στοκμόλης, Μα είπαν νομίζω να έχουν κανένα πρόβλημα με τη δεκαετία τη Πολωνία, έχουμε κάτι τέτοιο ήδη. Είχαμε το Ταντιντάτ. Έχουμε το καντιντάτ που είναι σαν μπάτσελορ. Και γι' αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην αποδοχή του διπλώματος bachelor από τους βιομηχανικούς και οικονομικούς κύκλους. Εκείνοι που μας είπαν να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της Πολώνιας δεν κατάφεραν να αποφασίσουν πού εντάσσουν τώρα τα διπλώματα bachelor. Δεν το καταφέρουν αυτό. Πολλά πρέπει λοιπόν να γίνουν ακόμα. Και αν μας βοηθήσει η Κομισιόν και μας είπε ότι θέλει να το κάνει, γιατί χωρίς τη βοήθειά της δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία των bachelor. Και κατά δεύτερον, θα να ευχαριστήσω στους συναδέλφους που το έδειξαν. Η κυρία Καμερέβερ, παραδείγματος χάρη, το πρόβλημα της ε, συχνότητας της πολιτικής αυτής, γιατί είχαμε μια ανακοίνωση από την κυρία Γκρός, είχαμε μια συζήτηση με την κυρία Επίτροπο κλπ. Και τρόμαξε η κυρία Γκρός όταν της ρώτησα πού υπάρχει η πολιτική, η, ο πολιτισμός στην ε, πολιτική που προτείνεται. Γιατί λέγεται κάπου οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τομείς θα ληφθούν εξίσου υπόψη. Δεν τρέχει τίποτα. Πολιτισμός εκτός. Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν να μην καλύψουμε όλες τις πτυχές και στο τέλος να μην υπάρχει καμία δυνατότητα να έχουν καλυφθεί όλες οι συχνότητες δηλαδή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και πολιτικά και πολιτισμικά και θα ήθελα να συζητήσετε το θέμα αυτό με την κυρία Κρόση. Η κυρία Κρόση με κάλεσε για καφέ και θα προσπαθήσω να το συζητήσω σοβαρά τη. Αντί να βάλουμε γάστρα στο καφέ, θα βάλουμε τα σημαντικά αυτά θέματα στο καφέ μας. Κάτι άλλο που ξεκίνησε αυτή η Επιτροπή εδώ τον Ιούνιο. Είχαμε μια διάσκεψη, ένα συμπόσιο αν θέλετε, για το θέμα του πολιτισμού στην υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων και από το συμπόσιο αυτό που είχαμε με την ΟΝΙΚ και με άλλους ξεκινήσαμε να, ε, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τώρα μία ε, έκθεση πρωτοβουλίας για το θέμα η κυρία Σάκε την ανέλαβε και ελπίζω να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα μπορείτε να συζητήσετε και με την Ριάστον. Εγώ συζήτησα με τον κύριο Έλμα Μπρόκ που προωθεί αυτές τις σχέσεις και στείλαμε από κοινού μια επιστολή στην κυρία Έσο, μπορώ να σας την ε, μεταβιβάσω, που είπαμε ότι θα πρέπει σε εξωτερικές σχέσεις να παίζει σημαντικό ρόλο και ο πολιτισμός. Είναι ένα από τα εξωτερικά μας προϊόντα. Βρισκόμαστε λοιπόν στη σωστή άκουσα και θα ήθελα να σας υποστηρίξουμε. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ αγαπητή κυρία Επίτροπε. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους επόμενους δύσκολους μήνες και ελπίζω ότι θα σας δούμε το αργότατο τον Γενάρη. Εδώ ίσως και το Δεκέμβριο, Άρα τι θα γίνει εδώ μεταξύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Πριν περάσω στο επόμενο σημείο, θα ήθελα να σας πω κάτι ακόμα. Αύριο έχουμε την ακρόση για τον κινηματογράφο. Δυστυχώς. Αυτό το πόστερ που θέλαμε να προετοιμάσουμε δεν είναι πολύ καλό τελικά. Είναι όλο μαύρο, μετά κάπου αναφέρεται το θέμα ε, και κάπου λέει Doris Pack. Κανένα δεν θα έρθει ούτε για τη μαυρίλα που υπάρχει, ούτε για το όνομα Doris Pack. Έχουμε δημιουργού από την Πολωνία, από την Ιταλία. Κανένα δεν αναγράφεται εκεί. Η γραμματεία δεν είναι υπεύθυνη από ό,τι μα είπαν. Άλλοι τα κάνανε έτσι. Αυτό είναι μη πολιτιστικό αν θέλω να το πω έτσι. Ωραία. Έβγαλα το άχτι μου τώρα που σας το είπα. Σας παρακαλώ αύριο να φέρετε όσους συναδέλφους μπορείτε ε, στην ακρόαση αυτή. Έχουμε πολύ σημαντικούς ε, δημιουργούς κινηματογράφου. Πρέπει με την παρουσία μας να δείξουμε ότι ενδιαφερόμαστε για όλα αυτά και ότι λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη αυτά που λέμε για το ψηφιακό κινηματογράφο. Αύριο λοιπόν μετά ψηφοφορία καλό να παραμείνετε, μην εξαφανιστείτε. Ναι, στην ψηφοφορία είναι συνήθω όλοι παρόντε. και σα παρακαλώ τι επόμενε δύο ώρε μετά την ψηφοφορία να μην βάλετε τίποτα άλλο στην ατζέντα γιατί έχουμε πάρα πολύ έντονη παρουσία από τη βιομηχανία κινηματογράφου. Ωραία. Τώρα στο σημείο 5. Έχουμε καλέσει του διοικητέ του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομάγνου για την νεολαία. Όσοι δεν ξέρετε, δεν θέλω να σα πω. Ε, λίγο φω αφήστε, ε. Μην τα σκοτειάσετε τελείως. Λοιπόν, ε, θα ήθελα να σα πω ότι πρόκειται για μια ιδέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είχε ξεκινήσει τότε από τον πρόεδρο Πέτερινγκ και από τους οργανωτές του βραβείου ΚΑΛ που υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Από εκεί ξεκίνησε. Αυτό το βραβείο δίνεται σε νέους μεταξύ 16 και 30 που προωθούν ε, μια κατανόηση των ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων. Είναι πολύ καλό βέβαια ε, εκείνοι που συμπεριλαμβάνουν στις στρατιωτικό πάνω από ε, μια χώρα. Είχαμε 216 σχέδια από τις 27 χώρες μέλη που υποβλήθηκαν και εξολογήθηκαν σε δύο φάσεις. Η πρώτη ήταν στις τι χώρες υπήρχε μια επιτροπή επιλογής από δύο βουλευτές και ένα νεκρό πρόσωπο των Εθνικών Οργανώσεων Νεολαίας. Έγινε μια πρώτη επιλογή, μετά τα 27 αυτά εθνικά σχέδια υποβλήθηκαν σε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου συμμετείχε ο πρόεδρος Μπούζεκ, τρεις ευρωβουλευτές και τέσσερις εκπρόσωποι από το βραβείο ΚΑΣ από το Άχεν. Αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εξέλεξε. Το τρίτο βραβείο 2.000 ευρώ δόθηκε σε έναν Βούλγαρο όπου μηχανικοί από τρεις χώρες ε, δημιούργησαν ένα ρομπότ που, που χρησιμοποιεί ε, περιβαλλοντικές πηγές ενέργειας. Μετά είχαμε το δεύτερο βιβλίο 3.000 ευρώ για ένα Ιρλανδικό, Ιρλανδικό κύριε Κέλλη. Ένα σχέδιο βιβλίου για νέους ε, και το πρώτο βραβείο εδόθη 5.000 ευρώ σε ένα γερμανικό σχέδιο που λέγεται το τρένο της Ευρώπης και ένωσε 1500 μαθητευόμενους από διάφορα σχολεία για να δημιουργήσουν ένα τρένο ε, με, όπου και ο, η μηχανή και τα βαγόνια είχαν κατασκευαστεί σε διαφορετικές χώρες. Περίεργο. Λοιπόν, εμείς έχουμε τον εκπρόσωπο από τη Βουλγαρία, Μαρία Κότοβα από την Ελλανδία, Λάιν Μάτσιν Σίμενστατ και έχουμε τους, το γερμανό εκπρόσωπο Ζάσα Έμρεχ. Και θα σας παρακαλώ ρουσιάστε στα γρήγορα το θέμα του. Η κυρία Κότοβα πρώτα. Are you sitting here? Fine. Please. Start. The project. Good afternoon to everybody. Καλησπέρα σε όλους σας. Θα μιλήσω αγγλικά. Πρώτα απ' όλα να σας συστηθώ. Είναι το όνομά μου Μαρία Κότιβα. Ε, συμμετέχω δύο χρόνια τώρα στο BEST. Θα σας πω ότι είναι το BEST στη συνέχεια. Ε, ασχολούμαι με τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και εκπροσωπώ αυτό το βουλγαρικό πρότυπο που κέρδισε το βραβείο Κάρλο Μάγνου για φέτος. Ε, η παρουσίασή μου λοιπόν θα περιλαμβάνει τα εξή. Πρώτα απ' όλα θα σας πω τι είναι το BEST, αποστολή, όραμα, υπηρεσίες. Μετά θα πάμε πιο τοπικά στο BEST της Σόφιας. Μετά θα σας μιλήσω για τον ε, διαγωνισμό για μηχανολόγους ε, και ποιο ήταν το follow-up του βραβείου που πήραμε και έχουμε λίγο χρόνο για ε, ερωτήσεις και απαντήσεις. Λοιπόν, το Best Many Board of European Students of Technology. Ε, Συμβουλίο Ευρωπαίων Φοιτητών για την Τεχνολογία. Είμαστε μη πολιτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εργαζόμαστε εθελοντικά και στην Ευρώπη ε, από το 1989, την σημαντική αυτή χρονιά, εκπροσωπούμε τα τεχνολογικά ιδρύματα ε, και προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε ε, καταλαβαίνοντας καλύτερα τις διάφορες κουλτούρες και το διεθνές περιβάλλον. Γινόμαστε όλο και μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι. Εκπροσωπούμε αυτή τη στιγμή 86 ε, τεχνικά πανεπιστήμια, πολυτεχνία αν θέλετε, σε 30 ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε σχεδόν 3.000 ενεργά μέλη και οι υπηρεσίες μας φτάνουν περίπου το 1 εκατομμύριο φοιτητές. Το, το όραμά μας είναι η πολιτιστική ε, πολυμορφία. Ε, προσπαθούμε να ε, παροτρύνουμε τους φοιτητές να δρουν υπεύθυνα. Οι δραστηριότητες μας ενθαρρύνονται από το βασικό μας στόχο που είναι να φέρουμε κοντά τα τρεις κορυφές αυτού του τριγώνου πανεπιστήμια, δηλαδή εταιρείε και φοιτητέ. Ε, επίσης, ε, ε, προσφέρουμε σημαντική προστιθέμενη αξία στην εκπαίδευση που παρέχουν τα πανεπιστήμια. Αυτό το επιτυχάνουμε οργανώνοντας κάθε χρόνο πολλά ακαδημαϊκά σεμινάρια καθώς και ε, διαγωνισμούς μεταξύ μηχανολόγων. Αυξάνουμε τη συμμετοχή των ε, φοιτητών μέσω διαφόρων εκδηλώσεων ε, καθώς επίσης αυξάνουμε την ευαισθητοποίησή τους για τα θέματα αυτά. Επίσης βελτιώνουμε την εκπαίδευσή τους με άμεση εμπλοκή τους στα διάφορα θέματα. Φυσικά ένας καλός χώρος εργασίας είναι τελικά αυτό που έχει σημασία και γι' αυτό βοηθάμε τους φοιτητές μας με διεθνείς ε, πλατφόρμες ε, σταδιοδρομίας, υποστήριξη σταδιοδρομίας, διεθνείς εκθέσεις ε, σταδιοδρομίας κλπ. Για το Best Sofia, πριν από ένα μήνα γιορτάσαμε τα 10 χρόνια του θεσμού αυτού. Συμμετέχουν 35 ενθουσιώδεις φοιτητές σε εθελοντική βάση βεβαίω, που προσπαθούν να προωθήσουν την Ευρώπη και τις αξίες της μεταξύ των φοιτητών. Κάθε χρόνο οργανώνουμε ε, ακαδημαϊκά ε, σεμινάρια ή διαγωνισμούς ε, και άλλες εκδηλώσεις που σχετίζονται με τα μέλη του BEST. Τώρα σχετικά με το project, το δικό μας, Οργανώθηκε αυτό τον Οκτώβριο του 2009 ε, με συμμετοχή 15 φοιτητών από 15 διαφορετικές χώρες, χωρίστηκαν σε 5 ομάδες και εργάστηκαν ε, σε δύο βασικά έργα. Ήταν ο βασικός στόχος να ε, φτιάξουν ένα ρομπότ που ακολουθούσε κάποια απορία με αισθητήρε. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Το background αυτού του γεγονότος είναι το εξής. Θεωρούμε ότι οι φοιτητέ δεν έχουν πλήρη επίγνωση των πλεονεκτημάτων της συμπληρωματικής εκπαίδευσης και της ε, ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία. Και θέλαμε επίσης να τους δώσουμε την ευκαιρία να αναπτύξουν και να θέσουν σε πράξη τα, τις μηχανολογικές τους δεξιότητες και γνώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ θετικό. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν ε, αποτελεσματικά σε μια διεθνή ατμόσφαιρα και να επικοινωνήσουν, ούτως ώστε να έχουν μια καλύτερη κατανόηση της πολιτιστικής ε, πολυμορφίας και αυτό προωθεί τη μελλοντική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο διαγωνισμοί αφορούσαν μια case study και ένα team design. Στο case study ανέλαβαν ε, ένα έργο από μια ε, εταιρεία. Ανέλαβαν να σχεδιάσουν μια μηχανή, ένα μηχάνημα για ανακύκλωση. Και το team design, ο ομαδικός ε, σχεδιασμός, αφορούσε το σχεδιασμό του ρομπότ. Στο πλόκτη έγινε η εκδήλωση για το project αυτό, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, όπου οι συμμετέχοντες έμαθαν και για την ιστορία της Βουλγαρίας και τις παραδόσεις της. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βρεθούμε στην ε, ε τελετή απονομή στο Άχεν, γιατί είχαμε το πρόβλημα το, με την φεστιακή έκρηξη τον Μάιο όμως ήμασταν προσκεκλημένοι στο κέντρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στη Σόφια και πήραμε τα βραβεία μας και βλέπετε τα φωτογραφίες από την τελετή αυτή. Τι έγινε τώρα μετά την ε, ε, απονομή αυτού του βραβείου, όταν λάβαμε αυτό το βραβείο και μετά. Τέλη Αυγούστου οργανώσαμε μια εκδήλωση για την εκπαίδευση με συμμετοχή 21 διεθνών φοιτητών τεχνολογίας επιλέγησαν με βάση τα ε, επιστολές αιτιολόγηση που έστειλαν και μετά από συνεντεύξεις δημιουργήσαμε τρία θεματικά δίκτυα όπου συλλέγονταν τα αποτελέσματα αυτής της εκδήλωσης και προωθούνταν στους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα της εκπαίδευσης. Είχαμε και εκπροσώπους εταιριών στην εκδήλωση έγινε και μια συζήτηση σχετικά με το πώς μπορεί να γεβηρωθεί με επιτυχία το χάσμα ανάμεσα στα πανεπιστήμια και στην επαγγελματική ζωή. Οι συμμετέχοντες φοιτητές ήταν τελειόφοιτοι οι περισσότεροι οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων μπορούσαν να δώσουν μια πλήρη εικόνα λοιπόν. Ε, πρέπει να σας πω ότι θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το βραβείο αυτό που λάβαμε γιατί αμφιβάλαμε στην αρχή αν μπορούσαμε να οργανώσουμε κάτι τέτοιο και επίσης με την ε, υποστήριξη ε, του προγράμματος Youth in Action ε, πραγματοποιήσαμε ένα project συνεργασία Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Γαλλίας σχετικά με την φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με την Ιρλανδία. Παρακαλώ, ε, περάστε εδώ. Εδώ δίπλα στην ε, κυρία από τη Βουλγαρία. Λίνε Μάτσεν, Okay. Go. Γεια σας. full screen. Slideshow. Okay. Um, my name is uh, Line Εκπροσωπώ μια μικρή, ένα μικρό εκδοτικό οίκο που λέγεται Broken Demands Press. Είμαι δημοσιογράφος. Δεν είμαι Ιρλανδή. Είμαι Νορβηγή. Δεν είμαι καν, δηλαδή, υπήκος χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώ, το σχόλιο του Πρόεδρου ήταν εκτό μικροφώνου. Πήραμε το δεύτερο βραβείο με το βιβλίο You Are Here που βλέπετε το εξώφυλλό του στην πρώτη διαφάνεια. Πρόκειται για μια ανθολογία με συνεισφορές από 8 νεαρά άτομα από διάφορες χώρες της Ένωσης και το επιμελήθηκα εγώ και ο κύριος Χόλντεν που είναι Ιρλανδός εξού και το Ιρλανδικό σχέδιο. Όπως σας είπα, η Broken Demands Press είναι ένας μικρός εκδοτικός οίκος που ιδρύθηκε το 2009, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Μας ενδιαφέρει η λογοτεχνία, η πολιτική και οι καστικές τέχνες. Το βιβλίο αυτό λοιπόν, You Are Here, δεν ξέρω, εσείς διαβάζετε αυτά που γράφει διαφάνεια. Τέλος πάντων, στο δικό μου το κομπιούτερ είναι λίγο πιο αχ, ε, αχνό το πίσω. Ε, τώρα δεν φαίνονται καλά τα, τα γράμματα. Πάντως, κατ' ουσίαν πρόκειται, πολύ γενικά, για το να ζει κανεί στην Ευρώπη 20 χρόνια μετά την πτώση του τείχου του Βερολίνου. Τι θα πει δηλαδή να είναι κάποιο ε, νεαρός Ευρωπαίος ε, που θεωρεί δεδομένη την αδιέρετη Ευρώπη, την ενωμένη Ευρώπη. Η ιδέα ουσιαστικά ήταν δική μου και του άλλου επιμελητή, του Τζον Χόλντεν. Το 2009, μάλλον όχι, το 2008. Είμαστε στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης που χάθηκε ξαφνικά το αίσθημα της ε, εθνικότητας. Περιβαλλόμαστε από κόσμο που έκανε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που μπορεί να μην είχαν σχέση με την χώρα καταγωγής τους αλλά με την Ευρώπη συνολικά, γενικά. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η γενιά στην οποία ανήκουμε εγώ γεννήθηκα το 85, ο Τζον το 84. Ανήκουμε λοιπόν και δυο σε αυτή τη γενιά που δεν έζησε το τείχος του Βερολίνου. Και θέλαμε να δούμε ακριβώς ε, το ότι δεν έχουμε αυτό σημείο αναφοράς ε, ως γενιά. Θέλαμε να δούμε ακριβώς ε, πώς το ζούμε. Αυτή λοιπόν η γενιά στην οποία ανήκω, όλα τα προγράμματα Εράσμους και τα λοιπά, τις μετακινήσεις τις ελεύθερες, ε, τα θεωρούμε δεδομένο. Άρα όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε και από το ενδιαφέρον για τη δική μας γενιά, αλλά και από το ενδιαφέρον μας ε, για το καλλιτεχνικό πολιτιστικό έργο νεαρών Ευρωπαίων. Έτσι λοιπόν, γεννήθηκε η ιδέα αυτής της ανθολογίας. Να σας πω λίγα πράγματα για αυτό το project. Κάναμε αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Νεολαία ενδράση, Προσπαθήσαμε να βρούμε άτομα που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτή την ανθολογία και για κάποιους μήνες ουσιαστικά αυτό που κάναμε είναι να ψάχνουμε, να βρούμε ενδιαφέροντα άτομα για να τα συμπεριλάβουμε στην ανθολογία. Καταλήξαμε λοιπόν σε ένα μείγμα από φίλους, φίλους φίλων, άτομα, νεαρά τέλο πάντων και αυτό που θέλαμε ήταν να επεξεργαστούμε ακριβώς την ιδέα αυτή που σας είπα για την γενιά μας και πώς είναι να ζεις και να εργάζεσαι σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. ίσως ε, ω ανθολογία το βιβλίο να είναι μοναδικό στο είδο του. Υπό την έννοια ότι εμεί ω επιμελητές, ε, ω συντάκτε ε, θέλαμε και εμείς ε, να υπάρχει το στοιχείο τη έκπληξη. Αφήσαμε δηλαδή τα άτομα τα οποία έγραψαν να γράψουν αυτό που ήθελαν και θέλαμε να εκπλαγούμε και εμεί ουσιαστικά, να, να μην γνωρίζουμε εκ των προτέρων το αποτέλεσμα. Τα άτομα αυτά ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Θα, θα, θα μιλήσω συγκεκριμένα για αυτού, στη συνέχεια. βρήκαμε και αυτούς οι οποίοι θα φιλοτεχνούσαν και το, την εικονογράφηση, το σχεδιασμό. Θέλαμε να κάνουμε και εμείς ένα ωραίο βιβλίο και θέλαμε και από την εικονογράφηση ε, και το σχέδιο, την όλη, τον όλη παρουσίαση επειδή το βιβλίο γράφεται σε πέντε διαφορετικές γλώσσες, θέλαμε να τονίζει και το σχέδιο εικονογράφηση ακριβώς αυτό το, το στοιχείο, τον πολυγλω, την πολυγλωσία μεταξύ άλλων. Στις 10 Νοεμβρίου λοιπόν του 2009 ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή δηλαδή με την 20η επέτειο από την πτώση του του Βερολίνου, συνέπεσε σκοπίμος και έγινε στο Βερολίνο. Ακριβώς, για αυτό το λόγο. Στείλαμε το βιβλίο σε διάφορους ε, οργανισμούς πολιτικούς ε, και οικονομικούς ε, μετά την παρουσίαση αυτή. Τώρα, ε, είναι λίγο δύσκολο να μιλήσω για το βιβλίο, γιατί τα θέματα με τα οποία καταπιάνονται οι συγγραφείς είναι πολύ διαφορετικά το ένα με το άλλο. Θα μπορούσα να αναφέρω κάποια παραδείγματα βέβαια. Παραδείγματο χάρη υπάρχει ένα άρθρο για τους μετανάστες στο Βερολίνο. Τι περιοχές προτιμούν, πού κινούνται γενικώ οι μετανάστες. Υπάρχει ένα δοκίμιο το οποίο μιλάει για την ε, πολιτική ένταξης ε, στην Ιταλία για αυτά τα τείχη ουσιαστικά που χωρίζουν κάποιες κακόφημες, κάποιες κακές περιοχές ε, της πόλης από, την υπόλοιπη, από τις την υπόλοιπη πόλη. Υπάρχει επίσης ε, ένα θεατρικό έργο από δανό συγγραφέα. Υπάρχει ένα άρθρο για ένα πολιτικό ακτιβιστή από τη Λευκορωσία. Η εμπειρία συγκεκριμένα τη και αυτή από την καταπολέμηση τη δικτατορία. Και γενικώ έχουμε και δοκίμιο, έχουμε και υποκριτική, δηλαδή έχουμε θέατρο, έχουμε ποίηση, εικαστικές τέχνες, πέντε διαφορετικές συνεκλώσει, γερμανικά, πολωνικά, λευκορωσικά, δανεικά, αγγλικά και μεταφράστα στα αγγλικά βέβαια. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο ασχολείται με την Ευρώπη ακριβώς. Ε, θέλαμε πάντως να δείξουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι τα αγγλικά και γι' αυτό καταλήξαμε σε αυτό, το, το την πολύγλωση έκδοση. Και εδώ έχετε, έχετε ένα κατάλογο με αυτούς που έχουν συνεισφέρει σε αυτό το βιβλίο. Μάλλον δεν βλέπετε και τίποτα, αλλά τέλος πάντων. θα σας διαβάσω εγώ. Είναι η ευστριακή Πίτρια Αν Κότεν που ζει στο Βερολίνο, είναι η Άννα Μπρό που είναι σεναριογράφος θεατρικών έργων από τη Δανία, η Αγνιέσκα Τροτσκίεβιτς που είναι νοβελίστα, συγγραφέας, ο Μάρτιν Τζον Κάλαναν είναι εκαστικός από την Αγγλία, η Βόλια Μαρτινέγκα από τη Λευκορωσία, πολιτική ακτιβίστρια, η Φραντσέσκα Μουσιάνη, κοινωνιολόγος από την Ιταλία, αλλά που έχει την έδρα της στο Παρίσι, ο Κριστόφα Φανγκέρεβι που είναι συγγραφέας, κριτικός τέχνης και η Ούρσουλα Βόσνιακ που είναι κοινωνική ανθρωπολόγος. Γερμανίδα αλλά πολωνικής καταγωγής και οι επιμελητές, ε, οι συντάκτες, Τζον Χόλτεν Ιρλανδία και οι υποφαινομένοι. Λίνε Μάτστεν Σίμενσταντ. Επίση, θέλαμε το βιβλίο αυτό ουσιαστικά να είναι και ε, ένα ξεκίνημα για τον εκδοτικό μα οίκο που αναστεί νέα ταλέντα. Ένα από αυτά λοιπόν είναι η Ανκότεν. θα εκδώσουμε σύντομα μία συλλογή ποιημάτων από την Ανκότεν. Αυτό είναι το επόμενό μας ε, project δηλαδή. Αυτά, αυτά είχα να σας πω. Thank The... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίος ομιλητές, πρώτο βραβείο, ο κύριος Έμπος. Jetzt geht es um einen Schmalspurzug. Bitte. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εγώ θα κάνω την παρουσία μου στα γερμανικά. Πολύ ωραία λέει η πρόεδρος. Λέγομαι Στάζα Εμρίχ, εκπροσωπώ το σχέδιο ΣΕΝΣΕ, το τρένο για την Ευρώπη. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ευκαιρία να σας παρουσιάσω εδώ αυτό το σχέδιο. ΣΕΝΣΕ, τι σημαίνει αυτό? Computer Numerical Control σημαίνει. Δηλαδή προγραμματισμένη επεξεργασία από ε, μηχανές. Λοιπόν, πώς μας ήρθε η ιδέα. Το 2006 είχαμε μια προσπαθιαυτική συνάντηση στις 10 Νοεμβρίου συγκεκριμένα και αυτό που βλέπετε είναι τα αποτελέσματα, η πρώτη εικόνα αν θέλετε που είχαμε τότε. Πριν να περάσουμε στην εικόνα αυτή στον πίνακα δεν είχαμε καμία ιδέα, κανένα όραμα, αλλά ο επικεφαλής του σχεδίου άρχισε να ζωγραφίζει ένα τρένο και αυτό ήταν μετά αυτό στο οποίο καταλήξαμε. Το σχέδιο μας αποτελείται από 24 ε, σχολεία από 21 χώρες δηλαδή ορισμένε χώρε εκπροσωπούνται από περισσότερα του ενός σχολεία και προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να τις πείσουμε να συμμετάσχουν σε αυτό το σχέδιο. Και δημιουργήσαμε διάφορες ομάδε εργασία σε συναντήσει που είχαμε, κάθε μια ασχολείται με άλλο θέμα και κατασκεύαζε επίση αυτό που χρειαζόταν. κάθε χώρα έπρεπε να κατασκευάσει μόνη της το βαγόνι που εκπροσωπούσε κατά τον ιδανικότερο δυνατό τρόπο αυτή τη χώρα. Πέντε συναντήσεις είχαμε στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία και στο Βέλγιο. Από το 2006 μέχρι το 2009, 10. Εδώ βλέπετε θαυμάσια πώς εργαστήκαμε. Βλέπετε δύο Ισπανούς που συνεργάζονται με ένα Γερμανό και σκέφτονται τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την οργάνωση. Μετά βλέπετε πώς δημιουργούνται τα βαγόνια, το κάτω μέρος των βαγονιών με ψηφιακή τεχνολογία, πέντε χώρες που εκπροσωπούνται. Εδώ βλέπετε το μοντάζ της ε, μηχανής και η προσαρμογή της ε, σύνδεσης με τα βαγόνια. Μετά έχουμε εδώ μια συνάντηση από την τελευταία συνάντηση στο Bad Korotsnacht στη Γερμανία που είχαμε τη δοκιμαστική λειτουργία του τρένου αυτού και μετά από διάφορες βελτιώσεις πραγματικά το τρένο αυτό ξεκίνησε και έτσι μπορέσαμε να εφησυχάσουμε. Και εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια ταινία τώρα αλλά για τεχνικούς λόγους δεν λειτουργεί από ό,τι φαίνεται. Το 2009 τον Απρίλιο είχαμε ήδη τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε το τρένο μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε έρθει 50 άτομα περίπου που παρουσιάσαμε αυτό το τρένο στον χώρο Γεούδη Μελουίν και το καταπληκτικό μετά ήταν ότι κερδίσαμε το πρώτο βραβείο, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεολαίας Καρολμάγνου. Το 2001, 11 συγγνώμη, θα υπάρχει ένα άλλο σχέδιο συνέχειας πάλι ένα τρένο, αλλά θα αναπτύξουμε το δίκτυο ΣΕΝΣΕ, δηλαδή θα μισούς άλλες χώρες και δεν ξέρουμε αν θα συμμετάσχουν όλοι οι παλιοί μας εταίροι. Άρα θα προσπαθήσουμε να ε, εντάξουμε και άλλες, άλλες σχολεία από άλλες χώρες και τα βαγόνια αυτά θα έχουν ίσως σαν ε, το χαρακτηρικό σημείο κάποιες, ε, ε, κάποιους κανόνες της φυσικής. Και μετά έχουμε και κάτι άλλο. Θέλουμε να ενσωματώσουμε εκεί ένα European Electronic Map. Δηλαδή, δίπλα στις ράγες του τρένου θα υπάρχει ένας χάρτης της Ευρώπης και όταν το βαγόνι από την ελόγω χώρα περνάει από εκεί, τότε στο χάρτη θα βλέπουμε να φωτίζεται η χώρα από την οποία προέρχεται αυτό το βαγόνι. Δύο χρόνια θα πάρει αυτό πάλι. Κατά πέσα θα αρχίσουμε δε την 1η Αυγούστου 2011. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα και προηγουμένως, ζητούμε να βρούμε και άλλες, άλλα σχολεία εταίρους και από τις χώρες που είχαν συμμετάσχει μέχρι στιγμής ίσως και από άλλες χώρες. Ίσως να μπορέσουμε να εκπροσωπηθούν όλες οι χώρες τώρα πια. Αυτά. Εγώ εκπροσωπώ και το σχολείο που συνενώνει τα πράγματα, είναι η BBS, τη GHS, στο Bad Kreuznach στη Γερμανία. Εμείς, εάν ε, θέλετε δηλαδή να ε, να συμμετάσχετε, να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Παρακαλώ, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ ωραίες αυτές οι παρουσιάσεις. Είναι πολύ ευχάριστο να ακούει αυτό, κανείς αυτά τα πράγματα και να δει πώς οι νέοι ε, εργάζονται για την συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν οι συνάδελφοι έχουν ερωτήσει, παρακαλώ να τι υποβάλουν τώρα. Κατά τα άλλα, θα ήθελα να μεταβιβάσω την παράκληση του νεαρού συναδέλφου Εμρίχη αν υπάρχουν σχολές τέτοιου τύπου στις εκλογικές σας περιφέρειες να τους πείστε να συμμετάσχουν. Ερωτήσεις? Α, μάλιστα, μάλιστα. Η κυρία Κάμερεβερτ. Όχι, δεν έχω μια ερώτηση, μια παρατήρηση είχα την τιμή και την ικανοποίηση να συμμετάσχω στο, στη Γερμανική ε, Επιτροπή για το βραβείο αυτό και ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό να δει κανένα πόσο διαφορετικά σχέδια υπευρύθησαν, πόσο διαφορετικές ιδέες υπήρχαν. Φαντάζομαι και σε άλλες χώρες το ίδιο θα ήταν, όπως και στη Γερμανία. Και μου φαίνεται πραγματικά λυπηρό ότι αυτά δεν ακούγονται καθόλου. Κανένα δεν ξέρει το βραβείο αυτό εγώ πριν έρθω στο κοινοβούλιο δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα και νομίζω πραγματικά ότι είναι πολύ μικρή η δημοσιότητα αυτών των δραστηριοτήτων και στα ίδια τα κρατη και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε αυτά τα καταπληκτικά σχέδια ε, όχι μόνο για τους νικητές που έχουν καταπληκτικά σχέδια αλλά υπήρχαν τόσο καλές ιδέες που θα ήθελα να είναι καλύτερα γνωστές, να γίνουν καλύτερα γνωστές για να πείσουν έτσι ίσως ε, προς μέσα στα πλαίσια κάποιων προβλημάτων βελτίστων πρακτικών. Πώς θα μπορέσουμε έτσι να προωθήσουμε δημοσιότητα και εδώ και στα κρατημέλη. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα να μην είναι γνωστό Ποιε είναι αυτές οι καταπληκτικές ε, πρωτοβουλίες που υιοθετούν οι νέοι. Γιατί στο κάτω-κάτω αυτή είναι το μέλλον μας, αυτή και η Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα τα συγχαρητήριά μου στους τρεις ε, ε νέους που παρουσίασαν ε, αυτά τα έργα απόψε. Ε, νομίζω ότι είμαστε πολύ περήφανοι και ιδιαίτερα εγώ είμαι περήφανος που βλέπω για κάτι καλό να προέρχεται από τη χώρα μου. Ευχαριστώ τον Τζον. Δεύτερον, όντως θα πρέπει να γίνει πιο γνωστό ε, το βραβείο αυτό. Και πρέπει να συζητήσουμε τρόπους στο μέλλον ώστε οι άνθρωποι γενικά να το εκτιμήσουν περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος ε, Μπόρις. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια σε όλους τους ε, βραβευμένους είναι, θα άξιζε οι καλές αυτές πρακτικές να μεταφραστούν σε κάτι ε, το πιο συγκεκριμένο. Η συνεργασία ανάμεσα στις ε, σχολές και στους εκδοτικούς οίκους. Παραδείγματος χάρη, επίσης το Κομένιους, πώς ε, κάτι που υπάρχει μπορεί να αξιοποιηθεί με βάση αυτές τις ε, νέες ιδέες. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω την Πρόεδρο αν μπορούμε να έχουμε κι εμείς αυτό το βιβλίο. Ε, που μιλάει για την ενσωμάτωση των νέων ε, Ευρωπαίων κλπ. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να το έχουμε και εμείς να το δούμε αυτό το βιβλίο. Μα το πέρσι είχαμε ζητήσει, είχαμε πει ε, ποιοι από τους συνεργάτες θέλουν να συμμετάσχουν. Αυτές οι ανακοινώσεις πολλές φορές δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη γιατί δεν ξέρει κανένα πόσο σοβαρά είναι. Τώρα ξέρουμε περί μας πρόκειται και ίσως γι' αυτό και θα μπορούσαμε να πάρουμε και την πρόταση της συναδέλφου Καμερέβερτ. Δηλαδή, είναι καλό να ξέρουμε ποια είναι τα παραδείγματα που βρίσκαν στα διάφορα κράτη. Γιατί οι συνάδελφοι, εμείς δηλαδή, δεν μπορούμε σε εκλογικέ μας περιφέρειες να τα προωθήσουμε τα σχέδια αυτά και από κοινού να κάνουμε μια παρουσίαση. Ποιες είναι οι ιδέες που έχουν οι νέοι, τι καταφέρνουν οι νέοι. Η Κία Καμπρέβερ ήταν παρουσιακή. δεν ξέρω από τη Γερμανία ποιο ήταν. Α, η Σαβίδα Φράιμ. Εντάξει. Ε, θα μπορούσαν να προτείνουν οι δύο κυρίες αυτές κάτι στην ε, Βορειοειρλανδία Βεσφαλία. Θα μπορούσαν να πούνε κάτι και στου συναδέλφου από τη Βαβαρία σου, να κάνουν και εκείνοι κάτι με του δικού του υποψήφου. Έτσι θα μπορέσουμε, ε, νομίζω, και οι νέοι που δεν κέρδισαν το βραβείο, όλοι εκείνοι που κατέβαλαν προσπάθειες να έχουν πιο ευρύ κοινό θα φροντίσω ακόμα, μια που ξέρω τη διαδικασία, να σα τη μεταβιβάσω. Ε, για σκέψω, να το θυμηθούμε αυτό, τη διαδικασία. Κυριακό και λέει Πώς τα Συμφωνώ με την πρόταση. Νομίζω ότι πρέπει να ε, αναλάβουμε να κάνουμε κάτι στις χώρες μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα πόρταλ ή κάπου που μπορεί να έχουν πρόσβαση όλοι και όπου μπορεί να δει κανεί ποιοι είναι οι νικητές και ποιοι είναι και αυτοί που δεν ε, κέρδισαν το βραβείο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό για κάθε κράτος. Ευχαριστώ. Μας, ε, πολλοί μας λένε, από σχολεία έρχονται σε επαφή, επαφή μαζί μας, μας λένε τι είναι η Ευρώπη, για την Ευρώπη θα ήταν καλό να τους πούμε ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο, γιατί θα πρέπει να το κοινοποιήσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Ωραία. Θα προφαντήσω να έχουμε ε, μια συνοψή του ότι υπάρχει αυτό, περί τίνος πρόκειται, πώς γίνεται και θα το στείλω στους συναδέλφους ούτω ώστε όλοι να ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο. Ένα αυτό. Και αν υπάρχει ένα πορτάλι κάτι στο διαδίκτυο, θα πούμε πού υπάρχει, πού μπορεί κανένα να δει τα σχέδια αυτά. Αλλά βέβαια θα πρέπει κανένα και να διαβάσει αυτά. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πάρα πολλά ε, email που παίρνουμε και πολλές φορές δεν ξέρουμε κατά πόσον όλα είναι σημαντικά. Ίσως κάτι θα μπορούμε να πούμε ότι είναι σημαντικό και για τη δική μας εργασία στις εκλογικές μας ε, περιφέρειας. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Κλείνουμε τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ τους ε, τρει συνεκητές. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και σπεριτέρω εργασία σας. Και να δούμε ποιο θα κερδίσει του χρόνου. Γιατί η ιδέα αυτή ξεκίνησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό και του χρόνου θα καλέσουμε τους νικητές. Δεν θα είσαστε εσεί κατά πάσα πιθανότητα. Πολύ θα πήγαινε αυτό αλλά ελπίζω ότι θα είστε ικανοποιημένοι να παίρνω το βραβείο και κάποια άλλη και θα συνεχίσετε στι εργασίε να έχετε κάποια συνέχεια. Γιατί είπατε εσεί ότι θέλετε περισσότερα βαγόνια, χρειαζόστε περισσότερου συνεργάτε και τα βαγόνια χρειαζόστε νέε τεχνικέ και τεχνολογίε. Πολύ ωραία αυτά όλα. Και εσεί θα έχετε οπωσδήποτε ένα νέο σχέδιο για το βιβλίο και εσεί στον τομέα σα, στη Βουλγαρία, θα φροντίσετε οπωσδήποτε η, η τεχνική εκεί και η μηχανική να έχουν νέες εφευρέσεις για να είναι καθαροι ε, το περιβάλλον μας ή να καθαρίσει. Ωραία. Περνάμε στους μία εξημείρες της διάταξης. Εγώ είμαι η συγγήτρια. Πρόκειται μια μήνες της διαταξης εγω ειμαι η Τώρα για συμμετοχη της ελβετιας στο πρόγραμμα Νεολαία Δράση και στο πρόγραμμα Δράση στον τομέα της βάθησης. Η Ελβετία πάντα ενδιαφέρεται για τον τομέα της ε, ε, εκπαίδευσης επαγγελματικής κατάρτισης νεολαία τον Αύγουστο 2009 επετέχθη συμφωνία με την Ελβετία για τη συμμετοχή της Ελβετίας στα δύο προγράμματα αυτά για την νεολαία και για την επαγγελματική κατάρτιση υπάρχει το άρθρο 216 σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να επικαιρώσει, να συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθεί η συμφωνία σε ισχύ. Δεν πρόκειται να ανοιχτούμε τη συμμετοχή μα. Εμεί χαιρόμαστε που συμμετέχει η Ελβετία σε πολλά πράγματα. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να τροποποιήσει τη συμφωνία ούτε το σχέδιο απόφαση. Έχει τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί, να το απορρίψει όμω. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο λόγο να το απορρίψουμε γιατί ε, πρώτον δεν μας κοστίζει τίποτα, η Ελβετία θα συμβάλλει οικονομικά στο πρόγραμμα αυτά και από την άλλη μεριά μπορούμε να χαιρόμαστε ότι διευρύνουμε τον ορίζοντά μας συμπεριλαμβάνοντας και την Ελβετία. Αξίζει αυτό. Τα κύρια στοιχεία τη συμφωνία είναι σχέδια και πρωτοβουλίε που βάλουν από συμμετέχοντα στην Ελβετία υπάρχουν τι ίδιε προποθέσει, κανόνε και διαδικασίε που ισχύουν τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, η Ελβετία θα δημιουργήσει μια εθνική υπηρεσία για το συντονισμό της εφαρμογής των προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο, όπως γίνεται και στις δικές μας χώρες, και θα καταβάλει ετήσια συνεισφορά και οι εκπρόσωποι της ε, Ελβετίας θα συμμετέχουν στη συνεδρίαση των επιτροπών ε, των προγραμμάτων ως ε, παρατηρητές εφόσον αφορούν την Ελβετία τα θέματα αυτά. Πρόκειται για το Νεολαία σε δράση και το πρόγραμμα δράσης για τη διαβίου μάθηση. Δεν μπορούμε νομίζω να είμαστε αντίθετοι. Διαφωνεί κανένας? Όχι. Στις 18 Νοεμβρίου λοιπόν επίσημα θα ψηφίσουμε πάνω στο θέμα αυτό. Τώρα κλείνουμε το σημείο 6 και περνάμε στο σημείο 7. Ευρώπη ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, ένα νέο πλαίσιο πολιτική για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Η εισηγήτρια μα είναι η κυρία Ράνερ. Είχαμε ήδη μια ανεπίσημη συζήτηση την περασμένη φορά. Θα ήθελα να σα δώσω τώρα το λόγο. Μέχρι τι 9 Νοεμβρίου 12 το μεσημέρι θα μπορέσουμε να υποβάλουμε τροπολογίε. Και στι 2 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε την πρόταση αυτή. Παρακαλώ κύριε Ράνερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, χαίρομαι που μπορώ να σας υποβάλω μια νέα πρόταση για τη γνωμοδότηση αυτή. Ε, πρέπει να εργαστούμε εδώ στενά με την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και ελπίζω τελικά οι ιδέες μας που αναπτύσσουμε εδώ να ληφθούν υπόψη στην Επιτροπή αυτή Μεταφορών με την οποία υπάρχουν κάποιες επαφές. μέχρι στιγμή ο τουρισμός δεν ήταν ένα θέμα που να απασχόλησε πολύ ούτε εμά ούτε την Επιτροπή Μεταφορών. Και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο για μας ότι ο τουρισμός είναι σημαντικός και για την απασχόληση και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και αυτό οδηγεί και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ο τουρισμός ήταν, είναι και θα είναι ένας κινητήρας της οικονομίας έχει όμως αντιμετωπίσει έντονες προκλήσεις. Αυτό που ενδιαφέρει εμένα είναι η γύρανση του πληθυσμού. Είμαστε όσο πάει και πιο ευκίνητοι αν θέλετε αλλά και πιο ε, μεγάλη στην ηλικία. Αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης είναι η εφορία και η προστασία του περιβάλλοντος και επίσης θα πρέπει η ζήτηση να τεθεί στα σωστά πλαίσια. Εγώ προσπάθησα να προετοιμάσω κάποιες ε, προτάσεις και χαίρομαι να λάβω τις δικές σας τροπολογίες γιατί αυτό θα σημαίνει ότι έχουμε τελικά ένα κείμενο που προέρχεται από το σύνολο της ε, Επιτροπής Πολιτισμών. Έχω βλέπω ότι τα ταξίδια ε, γίνονται όσο πάει και περισσότερο δημοφιλή. Και γι' αυτό καλούνται τα κράτη-μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να επιδείξουν ευληγησία σχετικά και να προσαρμοστούν στους νέους τύπους καταναλωτών και να λάβουν υπόψη νέε μορφέ τουρισμού, τι είπα. Ε, άτομα πιο ηλικιωμένα που έχουν ε, διαφορετικέ ανάγκε ή άτομα με ειδικέ ανάγκε. Γιατί όταν είναι κανένα ε, κάπω μεγάλο στην ηλικία δεν μπορεί να ανεβεί 150 σκαλιά για να δει το καμπαναριό τη εκκλησία κλπ. Η ζήτηση καθορίζει βέβαια και την ε, προσφορά και είπαμε ότι έχουμε εδώ να αντιμετωπίσουμε δημογραφικές μεταβολές που θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας. Το 2020 το 20% του πληθυσμού θα είναι πάνω από τα 65. Αυτό είναι μία όθηση για να μελετήσουμε το θέμα και να δούμε τι γίνεται με του εκείνου που έχουν παραμείνει νέοι, για να το πω έτσι, και όχι οι, οι, οι Τι θέλουνε, θέλουν να ταξιδέψουν με το λεωφορείο ή το φόβο να πετάξουν, θέλουν να κινηθούν με το δικό τους αυτοκίνητο. Υπάρχουν διάφορε κατευθύνσει. όπου υπάρχουν διαφορετικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντικό το προσωπικό που ασχολείται με τον τουρισμό και με το ότι θα πρέπει να είναι καλά καταρτισμένο το προσωπικό αυτό. Τονίζω γι' αυτό ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των προγραμμάτων όπως το da Νταβίντσι για την κινητικότητα των ε, φοιτητών ε, μέσα στα πλαίσια του Εράσμους παραδείγματος χάρη. Είναι αυτονόητο αυτό την Αυστρία ξέρω ότι κανένας δεν μπορεί να έχει μια θέση ε, στον τουρισμό αν δεν έχει εργαστεί και στο εξωτερικό. Ωραία. Αλλά θα πρέπει να το προωθήσουμε εμείς από την ευρωπαϊκή πλευρά γιατί μόνο αν ο επισκέπτης αισθάνεται σαν στο σπίτι του θα ξανάρθει. Αυτό είναι θέμα και επικοινωνία. Μεταξύ του προσωπικού καταρχήν και του επισκέπτη, του τουρίστ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προωθούν οι διεθνεί ανταλλαγές σπουδαστών από σχολεία επαγγελματική κατάρτιση, ούτω ώστε μεταξύ άλλων να βελτιώσουν τι γλωσσικέ του γνώσεις. Δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο να ακούει κανένα. Ε, σε πολύ σπασμένα οτιδήποτε πια δεύτερη γλώσσα, αν θέλει κανένα το αυγό να του το βράσουν 3 ή 5 λεπτά. Δεν του αρέσει και πάρα πολύ. Ε, βέβαια μπορεί κανένας να έχει μια εξειδίκευση, αλλά πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο να κατανοείται καλά ο επισκέπτης και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα στα διτά εκπαιδευτικά συστήματα που συνδυάζει τη μάθηση επιχείρηση με τη μάθηση σχολεία επαγγελματική κατάρτιση, αυξάνοντα έτσι τι επιδεξιότητε τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Αυτό υπάρχει στην Αυστρία ήδη. Τρει μήνε το χρόνο αποστέλλονται οι μαθητευόμενοι αυτοί από τι επιχειρήσει στη σχολή και τα αναπαλή. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε όλε τι χώρε. Οπωσδήποτε ο τουρισμό απαιτεί την συνεργασία μεταξύ των ε, επιχειρήσεων στου στόχους αλλά και των ε, τοπικών, ε, περιφερειακών και εθνικών οργανώσεων. Άρα και την δικτύωση των σχολείων. Ακριβώς στον τομέα του πληθυσμού. Το 10% των μαθητών αυτή τη στιγμή ε, στην Αυστρία βρίσκονται μέσα στα πλαίσια των επαγγελμάτων πληθυσμού. Δεν ξέρω για τις άλλες χώρες τι γίνεται. Πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό όμως. Δεν μπορούμε να αποκρύψουμε τη σημασία αυτών. Πάρα πολύ σημαντικό και γνωστό σε όλες είναι ε, πρωτοβουλίες όπως η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, το σήμα της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η διαδρομή του Σουηδρού Παραπετάσματος. Όλα αυτά μπορούμε να προωθήσουμε ως τμήματα της Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς. Θα πρέπει να θεωρούμε την Ευρώπη σαν ένα σφαιρικό στόχο για επισκέπτες από τρίτες χώρες. θα χρειάζεται βέβαια και το σχετικό μάρκετινγκ και γι' αυτό χαιρετίζω μια πολιτική όπως των προγραμμάτων EDEN που είναι γνωστά θα μπορούν να είναι και πιο, και πιο γνωστά γιατί το EDEN έχει τον εξή στόχο την προώθηση στόχων τουριστικών που δεν είναι τόσο γνωστά η μείωση της υπερπλήρωσης ορισμένων άλλων στόχων και νέο προσανατολισμό των ε, ροών τουρισμού σε, πιο παραδοσ... σε πιο λιγότερο παραδοσιακά μέρη, σε παραδοσιακούς στόχους. Μέχρι στιγμής έχουν δημοσιευτεί δύο εκδοχές. Στην Αυστρία πραγματικά ε, υπήρχαν περιοχές που ούτε και εγώ τις ήξερα και όπως γνώρισα. Μετά έχουμε το θέμα τουρισμός και αθλητισμός. Αναφέρθηκε ήδη σήμερα. Ξέρουμε πως μπορεί ο αθλητισμός να συμβάλλει στο ότι οι άνθρωποι να είναι πιο ικανοποιημένοι, εντό αγωγικών ευτυχισμένοι. Εδώ αναφερόμαστε στον βιώσιμο τουρισμό. Ακόμη και τώρα έχουμε τους ε, ειδικού εδώ για το ποδήλατο. Ξέρετε περί μας πρόκειται. Υπάρχουν ορισμένες μορφές ε, αθλητισμού που μπορεί ο καθένας να ασκήσει. Και άμα σκεφτεί κανένα πόσο μεγάλη ηλικία μπορούμε να γίνουμε σήμερα, βλέπουμε ότι ε, πολιτιστικές, τουριστικές εκδηλώσεις δεν γίνονται πάντα με τρόπο ούτως ώστε να μπορούμε να, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και μικρές ε, αθλητικές ε, εκδηλώσεις που δεν τις ξέρει ο καθένας και που μπορούν όμως να προσφέρουν κάποιες δυνατότητες. Πρέπει λοιπόν να γίνει καλύτερη διαχείριση των υφισταμένων ουσιακών προγραμμάτων με τη διάρκεια επαρκών χρηματοδοτικών πόρων για να επιτευχθεί η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Ποτέ δεν έχουμε βέβαια αρκετά χρήματα. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε και ανατομικοί και προγράμματα που υπάρχουν και μπορούν πραγματικά αξίζουν να υποστηριχτούν να το κάνουμε. Και τέλος, σας υπενθυμίζω ότι την περασμένη φορά συζητήσαμε ότι υπάρχει ο www.visiteurope.com που είναι μια πλατφόρμα που μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω κατά τη γνώμη μου. Παρουσιάζει όλα τα κράτη-μέλη και έχει σαν στόχο να αυξηθεί η προβολή της Ευρώπης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, παράγοντας πληροφορίες στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό επισήμων γλώσσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θυμάμαι παραδείγματος αυτό το αυστριακό βιβλίο που διατίθεται τώρα σε όλες τις γλώσσες πια. Αυτή η πλατφόρμα θα μπορούσε να είναι μια κομβική πλατφόρμα που θα συνδέει και άλλα προγράμματα και εφαρμογές. Εφόσον έχουμε μια τέτοιου τύπου πλατφόρμα θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Τελειώνω εδώ. Ντόρις, ξέρω, ανησυχείς. Τον Ιούλιο, Ιούνιο και τον Ιούλιο υπάρχει περισσότερο περισσότερος αλλά εγγνώση μου δεν το συμπερέλαβα αυτό στην έκθεσή μου. Δεν ξέρω, θα κάνω κι εγώ μία πρόταση. Εκείνοι που δεν εξαρτώνται από τις ε, σχολικές διακοπές ίσως θα μπορούσαν να ταξιδεύουν μέχρι και τον Οκτώβριο και από τον Απρίλιο μετά για να μην έχουμε μια συγκέντρωση στις συγκεκριμένες ε, εποχές. Αυτό είναι καλό και για τις επιχειρήσεις σχετικές αλλά και για τους επισκέπτες. Με χαρά περιμένω τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας και είμαι πεπισμένο ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μια καλή, καλή πρόταση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Η κυρία Κώστα έχει δει στο λόγο. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Συμφωνώ με πολλές από τις ε, υποδείξεις της και της απόψεις της. Νομίζω ότι πρέπει να μπορέσουμε να ε, ενισχύσουμε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να σας πω το εξής. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να δρομολογήσουμε αυτή τη γνωμοδότηση έχοντας στο μυαλό μας ότι ο πολιτισμός και ο ε, πολιτιστικός τουρισμός είναι, μάλλον ο πολιτιστικός τουρισμός είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του τουρισμού σήμερα στην Ευρώπη. Υπάρχει ένας νέος τρόπος ε, να βιώνει κανείς το ε, ευρωπαϊκό τουριστικό προϊόν μέσω αυτής της πτυχής. Διότι όπως είπαμε και σε άλλες συνεδριάσεις πιστεύω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ενώ έχουν αλλάξει πάρα πολύ σήμερα οι, τρόποι με τους οποίους βιώνει κανείς την τουριστική εμπειρία δεν είναι μόνο η επίσκεψη, δεν είναι μόνο μια εκδήλωση σημαίνει ε, το βίωμα ε, μιας ε, κατάστασης. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι η αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής για αυτό το θέμα είναι πολύ πιο σημαντική από ότι έχουν κατανεμηθεί αυτή τη στιγμή οι αρμοδιότητες ανάμεσα στις μεταφορές τρόποι μεταφορών κλπ. Και από την άλλη μεριά, το λόγο για τον οποίο έρχεται κανείς στην Ευρώπη. Δεύτερον, είναι σημαντικό να ε, υπενθυμίσουμε ότι παράλληλα με την πρωτοβουλία του σημείου 5 θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και να υπενθυμίσουμε ε, ακόμα μια φορά το πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους ευρωπαϊκές, τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές. Και τρίτον, ε, ανάμεσα στους τέσσερις άξονες της ε, υπάρχει ο βιώσιμος και υπεύθυνος τουρισμός. Νομίζω ότι και εδώ πρόκειται για μια ε, νέα ε, μορφή τουρισμού πέρα από τις εποχικές διακυμάνσεις με πολύ μεγάλη διαφοροποίηση και ε, με πολύ πιο έντονη συμμετοχή των περιφερειών στη διακυβέρνηση. Και επίσης υπάρχει και ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τις δημιουργικές πόλεις που αποτελούν ένα δίκτυο που μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και παράλληλα ε, με, το, με την πολύ σημαντική μνήμα που γίνεται σε κάποιες πρωτοβουλίες όπως για τις ευρωπαϊκές πολιτικές πρωτεύουσες θα έπρεπε να προωθηθεί περισσότερο ο πλούτος της Ευρώπης. Ένας τουρισμός δηλαδή που να βασίζεται σε μικρά κέντρα, σε μικρές κοινότητες της υπαίθρου ε, μικρών διαστάσεων. Και πιστεύω ότι από αυτή την άποψη θα πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα τη σύνδεση ανάμεσα στην προσφορά του πολιστικού τουρισμού και από την άλλη μεριά ε, σε μια πολιτιστική προσφορά προϊόντων, ε, ε, design κλπ. Πράγμα δηλαδή το οποίο προσφέρουν οι πόλεις και οι κοινότητες πέρα από τις κλασικές, τα κλασικά τουριστικά προϊόντα, ιστορία κλπ. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι υπάρχει μια διεύρυνση της προσφοράς που χάνει τον εποχιακό χαρακτήρα έτσι και απλώνεται ε, ευρύτερα. Ευχαριστώ. πολύ. Νομίζω ότι πραγματικά η παρουσία της γήτριας ε, ήταν πάρα πολύ εύστοχη. Ίσως ε, να θεωρείται η αρμόδια για τον τουρισμό η Επιτροπή Μεταφορών, αλλά νομίζω ότι η δική μας Επιτροπή ε, έχει ένα τεράστιο δυναμικό να βοηθήσει στην ανάπτυξη του τουρισμού ανά την Ευρώπη. Όπω είπε η συγγήτρια, ο πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, ο πνευματικό τουρισμό, ο αθλητικό τουρισμό είναι όλοι τομεί πολύ μεγάλη ανάπτυξη και δυναμικού, ιδίω αυτή τη χρονική στιγμή. Γιατί είναι... Και επίση πρέπει πάρα πολλά πράγματα να γίνουν για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον τουρισμό και να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο. Νομίζω ότι και οι νέοι έχουν δυνατότητες. Δεν θα πρέπει να τους ε, ξεχάσουμε. Όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το μείγμα. Νομίζω ότι τώρα έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τον τουρισμό, να αναπτύξουμε την οικονομία στην Ευρώπη και να δημιουργήσουμε μια αίσθηση ευρωπαϊκής ταυτότητας, για το οποίο άλλωστε συνέχεια συζητούμε. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια ταυτότητα ευρωπαϊκή στον τουρισμό που νομίζω ότι αν διαφημιστεί και προβληθεί σωστά θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριος Φίσας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω και εγώ ότι πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία, δηλαδή συνδυασμό τουρισμού και πολιτισμού. Θα ήθελα να τονίσω πάνω απ' όλα το ζήτημα της ενημέρωσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Μιλάμε για φεστιβάλ, μιλάμε για συναυλίες που μπορεί να είναι κάποια κονσέρτα κλασικής μουσικής αλλά μπορεί να είναι και συναυλίες για νέους. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν και η διαφήμιση, η προβολή Επίσης, οι διάφορες ομάδες ε, στόχοι, τα διάφορα τμήματα, είπαμε, ηλικιωμένοι, οικογενειακό τουρισμός, νεολαία, υπάρχουν διαφορετικά τμήματα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον τουρισμό με συγκεκριμένες ε, πολιτιστικές προσφορές στην προκειμένη περίπτωση. Και αν μιλήσουμε και για τον αθλητισμό, δεν έχουμε μόνο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, αλλά και η, πραγματικά η άσκηση, το να πάει κανείς να κάνει σκι στην Αυστρία ή να κολυμπήσει το καλοκαίρι στην Κώστα Ντελσόλ. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να προωθήσουμε και τον αθλητισμό για όλους. Υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα πάντα σε σχέση και με όσα λέγαμε πριν για τη νέα υπηρεσία εξωτερική δράση. Στην Ευρώπη έρχονται πάρα πολλοί τουρίστε από όλε τι υπήρου. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον οι τουρίστε αυτοί που δυνάμει θα έρθουν ε, στην Ευρώπη να έχουν ε, την κατάλληλη ενημέρωση ίσως και μέσω της εξωτερικής υπηρεσίας για την προώθηση του τουρισμού. Μπορούμε να προωθήσουμε σε αυτά τα πλαίσια και τον πολιτιστικό τουρισμό με τους νέους πρέσβεις, τις νέες πρεσβείες που θα έχουμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που μάλλον συμπεριέλαβε όλες τις πτυχές του τουρισμού. Ευχαριστώ πολύ, Χέλα. Έχουμε πολλά είδη τουρισμού και σε μεγάλο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκρίνεται στις ε, υφιστάμενες ανάγκες. Θα ήθελα όμως να αναφέρω δύο πράγματα. Την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διάσταση πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστώ που συμπεριλάβατε ορισμένα στοιχεία τα οποία υπερβαίνουν ε, το πλεονεκτήματα και τα προνόμια μιας χώρας. Νομίζω ότι πρέπει να προωθούμε ε, τις ευρωπαϊκές θεματικές ε, διαδρομές, παραδείγματος χάρη, σιδηρούν παραπέτασμα κτλ. κτλ. Η διαδρομή Σαντιάγο Δε Κομποστέλα. Κάτι το οποίο ίσως λείπει στην Επιτροπή Μεταφών και τη σχετική γνωμοδότηση είναι το εξής Σήμερα θα πρέπει να μπορούμε να επικοινωνούμε, να ταξιδεύουμε γρήγορα και αποτελεσματικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν είναι το θέμα των εταιριών των αεροπορικών low cost. Δεν διευκολύνει, μόνο, δεν μόνο αυτό τη μετακίνηση των τουριστών, αλλά και οι γρήγοροι σιδηρόδρομοι. Άρα και αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας πάντα στο πλαίσιο του τουρισμού. Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να υπογραμμίσω μια πτυχή που ανέφερε η συνάδελφος Ράνερ πολύ σωστά αλλά δεν το, τη βλέπω στη μετάφραση του κειμένου στα Ιταλικά η πτυχή δηλαδή του αθλητισμού σε σχέση με τον τουρισμό. Γιατί στην Ιταλία, και όχι μόνο στην Ιταλία νομίζω, όλο και περισσότερο ο αθλητισμός συσχετίζεται με τον τουρισμό. Μέσα από αθλητικές πρωτοβουλίες αναπτύσσεται μια γνώση ε, της τοπικής ε, κοινωνίας που αναπτύσσεται πάρα πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι πια πολύ νέοι και που συνδυάζουν αθλητισμό και τουρισμό. Κάτι που ε, ε, ε, αρχίζει να επικρατεί. Είναι κάτι το οποίο εντόπισε, ε, πώς το λένε, ανέφερε η ομιλήτρια στην παρουσίασή της, αλλά δεν το βλέπω στη μετάφραση στα Ιταλικά. Ευχαριστώ. Στο σημείο 5, δηλαδή, να μην αναφέρουμε μόνο αυτά που αναφέρονται, αλλά και οι πολιτιστικές διαδρομές γιατί θέλουμε στην ε, Ρωμανία παραδείγματος να έχουμε μια τέτοια διαδρομή. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και θα πρέπει νομίζω να ενταχθεί. Επίσης έχω προβλήματα με το δεύτερο σημείο. Έτσι πως έχει δεν λέει. λέει υπογραμμίζω ότι είναι σημαντικό να αυξηθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης με τη χρήση προγραμμάτων όπως το Λεωνάλο Νταμίτσι ε, για την κινητικότητα των ε, φοιτητών και τα βελτιώσουμε το Εράσμος για του επιχειρηματίες. Α μην έχουμε παντού ε, το Εράσμος και εμείς δεν έχουμε σαν στόχο να υποστηρίξουμε τους επιχειρηματίες. Εκείνοι πρέπει να επενδύσουν γιατί εκείνοι θα αφηληθούν με τις ε, τουριστικές δραστηριότητε. Θα σα βγάλω λοιπόν τους ε, επιχειρηματίες. Αυτό που ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να μαζέψει εμπειρίες στην διαμεθοριακή τομέα δεν είναι καλό επιχειρηματής και θα τον στηρίξω ούτω ή άλλω. Επίσης αυτές οι εμπειρίες στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ σημαντικέ για όλους εκείνους που δρούν στο τουριστικό τομέα και θα πρέπει να εκμεταλλευτούν όλα τα προγράμματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε οι ερευνητές ούτε το Εράσμου ταιριάζει εδώ. Κατά τα άλλα μου φαίνεται ότι είναι καλό και θα έλεγα όσον αφορά το Visit Europe δεν έχω κοιτάξει ποτέ μου ίσως να υπάρχουν κάποιες διαθυνδέσεις κάποια links για τα ευρωπαϊκά φεστιβάλ παραδείγματος χάρη. <coughs> Έχουν δική τους ε, πλατφόρμα. Αλλά άμα στο Visit Europe ε, λέει εκεί πηγαίνετε στην ε, πύλη για τα φεστιβάλ, καλό θα ήταν αυτό για όσοι ενδιαφέρονται για τα φεστιβάλ. Μπορεί κανένα να βελτιώσει και εγώ θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες. Θες κάτι να προσθέσεις, έλα. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω. Ε, σημείωσα κάποια πράγματα που ελέγχθησαν. Αυτό για το Visit Europe που θα μπορέσει να ενθαρρύνει κάποιε ε, περιφέρειες που δεν μπορούν από μόνος τους να τα καταφέρουν ε, για οικονομικού και άλλου λόγου. Για του επιχειρηματίε εντάξει, ναι, ναι, το σημείωσα αυτό, θα το βγάλουμε. Για τον ε, αθλητισμό, όπω είπε ο συνάδελφο Κορία, καυτό το θέμα για μένα και στι 10 Νοεμβρίου θα προσπαθήσουμε στο να δούμε τι γίνεται ε, ο θετισμός και Ευρώπη όπου έχουμε ένα παιχνίδι Ουγγαρία, όπου παίζουν η Ουγγαρία, η Σλοβία και η Κροατία ε, χόκι στον πάγο. Ναι, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούν να συνταθούν αυτά με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιο σχετισμό. Κατά τα άλλα βέβαια, ότι το αθλητισμός υπάρχει πέρα από τα σύνορα, εντάξει, ναι αλλά θα πρέπει να υπάρχει άμεσο χειρισμό με το θέμα του πολιτισμού και του τουρισμού. Οπωσδήποτε θα βρούμε κάποια δυνατότητα. Ωραία. Εδώ μπορώ να κλείσω αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να πάρετε όλα σας τα χαρτιά που θέλετε να πάρετε, γιατί αύριο είμαστε σε μια άλλη αίθουσα, σε ένα άλλο κτίριο. Πώς το είπαμε αυτό? Στο κτίριο Γιάν. 4Q1, 4Q1, αύριο το πρωί για την ψηφοφορία με τις κάρτες σας αν είναι δυνατόν παρακαλώ γιατί υπάρχουν ίσως διαφορετικές απόψεις που θα πρέπει να εντοπίσουμε. Λοιπόν, και να μείνετε και στην ακρόαση αύριο παρακαλώ. Λοιπόν, 10, 10 με μία αύριο. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Οι συντονιστές παρακαλώ να μείνουν στην αίθουσα. Okay können wir ganz schnell dafür sorgen, dass alle Nicht-Koordinatoren und Mitarbeiter den Raum verlassen. Παρακαλώ όσοι δεν είναι συντονιστές να φύγουν γρήγορα από την αίθουσα ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρία των συντονιστών. Herr Borgo ist neu im Ausschuss, hatte ich vergessen zu sagen.